Julian. So, good morning. Καλημέρα κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ καθίστε. Καλώς ήρθατε στη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων από τις Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Εξ ονόματος των συναδέλφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας πω ότι χαιρόμαστε που βλέπουμε τόσους πολλούς συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας και συμμετέχουν στην τελευταία αυτή διακοινοβουλευτική συνεδρίαση αυτής της θητείας και πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών ε, πριν από τις ευρωεκλογέ. Προτείναμε τρία θέματα που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε έναν απολογισμό της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής ε, και πολιτικής ασφάλειας και των μελλοντικών προκλήσεων. Πρώτα απ' όλα προτείνω να γίνει μια σύντομη συζήτηση μεταξύ μας για τα θέματα αυτά με εστιασμό για το πώς μπορεί να ενισχυθεί για το μέλλον πιθανώς με ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Στις 10 η ώρα μετά έχουμε τον Μισελ Μπαρνιέ για μια ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Brexit και ειδικά μετά τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις στην Βουλή των Κοινοτήτων Πρόκειται πολύ επικυρή συζήτηση και στις 11.30 θα έρθει ο Επίτροπος Ιωάννης Χάν για να συζητήσουμε μία από τις προτεραιότητες ε, της εξωτερικής πολιτικής, η ε, γειτονιά μας, ε, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και η διαπραγματεύση για τη Τέλος, θα έχουμε ένα γεύμα εργασίας όπου θα αναφερθώ στις μελλοντικέ μας εργασίες και συνεδριάσεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα με τη γενική συζήτηση για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Να σας μεθυμίσω ότι κάθε χρόνο το Συμβούλιο εγκρίνει μια έκθεση για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τις προτεραιότητες της ΚΕΠΑ για το επόμενο έτος. Κατόπιν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την δική του θέση με ένα ψήφισμα που προετοιμάζει η Επιτροπή μας πριν από λίγες εβδομάδες. Επίθυνα επιστολή σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια του ψηφίσματος, το οποίο εγκρίθηκε μεγάλη πλειοψηφία πέρυσι στις 12 Δεκεμβρίου. Στο ψήφισμα αυτό τονίζουμε μια σειρά προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, διερευνούμε πιθανού τρόπους για να προωθηθεί η ΚΕΠΑ. Παραδείγματο χάρη προτείνουμε την βελτίωση της λήψη αποφάσεων μέσω της σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ε, έχουν ζητήσει μεταξύ άλλων η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Μακρόν. Επίσης προτείνουμε να αντικατασταθεί η ομοφωνία στο Συμβούλιο για ζητήματα ΚΕΠΑ με ειδική πλειοψηφία. Αυτή είναι η τυπική διαδικασία για τις περισσότερες πολιτικές ένωσεις. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι η εξωτερική πολιτική είναι ιδιαίτερος ευαίσθητη και η πιθανή κατάργηση της ομοφωνίας ε, είναι ένα ζήτημα επίμαχο, αλλά θεωρώ ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να είναι μια παγκόσμια δύναμη μόνο εάν καταφέρουμε να απομακρυνθούμε από τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Θα ήθελα όμως να ακούσω και τις δικές σας απόψεις, ε, ειδικά των εθνικών κοινοβουλίων. Ένα άλλο θέμα, ε, στο οποίο συμφωνώ και εγώ και η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών, είναι ότι έχουμε ένα πιο απρόβλεπτο περιβάλλον ασφαλείας από ε, οποιαδήποτε άλλη εποχή από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη να διαφυλάξει την ασφαλειά της ε, και τα συμφέροντά της και τις αξίες της. Οπότε πρέπει να λάβει την μοίρα της ε, και να φερθεί ως μια πλήρως κυρίαρχη πολιτική και οικονομική δύναμη στις εθνείς σχέσεις να βοηθήσει να επιλύσει τι ε, διεθνείς συγκρούσει και να διαμορφώσει την παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτά από μένα. Τώρα προτείνω να χρησιμοποιήσουμε τα επόμενα 40 λεπτά για μια συζήτηση μεταξύ μας πριν έρθει ο κύριος ε, Μπαρνιέ. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πώς ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανταποκριθεί στι σημερινέ προκλήσει και θα θέλαμε να ακούσουμε πώς βλέπετε το όλο θέμα της ε, ειδική πλειοψηφία σε ζητήματα εξωτερικών, κάτι το οποίο φαντάζομαι θα παίξει ένα ρόλο και στην προεκλογική εκστρατεία. Για τα τεχνικά να ενημερώσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια ότι σας έχουμε δώσει κάρτες, ομιλίες, ε, σηκώστε τις για να ζητήσετε τον λόγο. Οι ευρωβουλευτές ζητούν τον λόγο ως συνήθως. Ορίστε. Α, έχουμε ήδη τον πρώτο μιλητή. Μάλιστα. Αυτά από μένα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Θα δώσω τον λόγο λοιπόν στον συνάδελφο και φίλο τον κύριο Κάνινς από την Λετωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σημαντική πτυχή της κοινή αμυντικής πολιτικής είναι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και μέχρι στιγμής ήταν πολύ επιτυχής. Οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορετικά σημεία επαφής. Η ανησυχία μου είναι η έλλειψη στήριξης ε, που βλέπουμε από την Ουάσιγκτον όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την συνεργασία με το ΝΑΤΟ μια που μιλάμε για τη ΣΥΠΑ. Και αν κάνουμε αρκετά για να επηρεάσουμε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις στην Ουάσιγκτον για να αναγνωρίσουν τις σημαντικές σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Μπορεί να μπορούμε να επηρεάσουμε τον Λευκό Οίκο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τα μέλη του Κογκρέσου, τα Think Tank, ακόμα και τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ για να τονίσουμε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Νομίζω θα ακούσουμε κάποιους συναδέλφους ε, και μετά ίσως μπορούμε να επανέλθουμε σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Με, τι θέτε να κάνουμε τώρα. Ένας και ένας μάλιστα. Οπότε τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Χάτζη Γεωργίου, Ευρωβουλευτής. Καλημέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ τους Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Να πω καταρχήν ότι δεν υπάρχει εδώ εκπρόσωπο του Εθνικού Κοινοβουλίου της Κύπρου και μερικά πράγματα από όσα θα πω αντικατοπτρίζουν τις θεσει και της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της Κύπρου. Γενικότερα ομω ξεκινώ από το, την τοποθέτηση πω η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στα παγκόσμια πράγματα δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει πιο θετικά παγκόσμιο ρόλο εάν καταφέρει πρώτα απ' όλα να λύσει προβλήματα του οίκου τη, Εάν ε, καταφέρουμε να αναπτύξουμε πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και αν καταφέρουμε τα κράτη-μέλη να αποδέχονται την κατανομή ε, μεταναστών ανάλογα με την δύναμη, την έκταση ή τον πληθυσμό τους. Να μην επιβαρύνονται δηλαδή μόνο κάποια κράτη. Και τρίτον, αλλά καθόλου τριτεύον, να λύσει οικονομικά προβλήματα των, πολιτών της. Ε, προβλήματα δημοκρατίας, ανάσχεσης ε, των ακροδεξιών λαϊκίστικων κινημάτων που φαίνεται ότι στις επόμενες ευρωεκλογές μπορεί να πάρουν περισσότερη δύναμη. Νομίζω λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε εσωτερικά για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ικανοί ε, στη δράση μας ε, στο, στο παγκόσμιο σκηνικό. Ε, έρχομαι τώρα στην ε, στο συζήτηση για την ειδική πλειοψηφία σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα καταρχήν προσωπικά υπάρχει ακόμα ασάφεια ε, για το για ποια θέματα μιλάμε ότι θα χρειάζεται αυτή η ειδική πλειοψηφία. Αν είναι για όλα δηλαδή ή αν είναι για κάποια συγκεκριμένα και πώς καθορίζονται αυτά τα συγκεκριμένα. Και εδώ τοποθετώ την θέση της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της Κύπρου. Η Κύπρος και νομίζω ότι και άλλα κράτη, μικρά ή νέα κράτη που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν, ανησυχούμε από την πιθανότητα οι αποφάσεις να παίρνονται με ειδική πλειοψηφία διότι αυτό θα συνεπάγεται αμέσως, ιδιαίτερα για μικρά κράτη, επαναλαμβάνω, ε, ότι ε, δεν μετέχουν των, των κοινών αποφάσεων. Ε, με αυτά σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Next on my list is Mr. Κατόπιν, κύριος Τσιγκάλης από την Λιθουανία. Yeah. Press red button. Ja, συνάδελφοι. Äh, ήθελα να τονίσω ότι σε αυτούς τους ε, ταραγμένους καιρούς ε, θα πρέπει να στηρίξουμε αυτήν την ε, γέφυρα με την άλλη Ατλαντικού και αυτό το οποίο είπε επίσης ο Λετωνός ε, συνάδελφος είναι σημαντικό. Η πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά της ε, διατλαντικής μας συμμαχίας η υπόθεση αυτή ε, με τα συνθήματα που αφορούν τον Τραμπ, ε, οι διαμάχες Μακρόν και Τραμπ, ε, είναι πράγματα που δεν χρειάζονται τώρα. Από τη δική μας τη σκοπιά η ασφάλειά μας βασίζεται στη φιλία μας με τον Καναδά, τη ΣΥΠΑ και την Αυστραλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτόν τον, αυτή τη συμμαχία του πολιτισμού και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κινηθούμε κατά αυτής της ε, συμμαχίας. Επίσης θα ήθελα να τονίσω, κύριε Μακάλιστερ, την απογοήτευσή μας όσον αφορά τις ε, σχέσεις μας ε, με το Συμβούλιο της ε, Ευρώπης. Γιατί έχουν αποκλειστεί δύο πρόσωπα από την Υπουργική Επιτροπή, δύο πρόσωπα που ήταν υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Κομπίλης, ε, ο οποίος δεν έγινε δεκτός ως υποψήφιος για Γενικούς Γραμματέας της ε, Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης. Μετά τα όσα συνέβησαν του τελευταίους δύο μήνες ε, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφοι τα τέσσερα κριτήρια. Γιατί ο Πρωθυπουργό ε, ήταν 8 χρόνια Πρωθυπουργό. Διατήρησε τη φιλελεύθερη γραμμή της χώρας μας σε καιρούς κρίσης. Είχαμε ζητήματα δημοσιονομικά και διατηρήσαμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη χώρα μας και είμαι πραγματικά απογοητευμένος για το ότι ο Πρωθυπουργό ε, δεν έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος ε, για την κοινοβουλευτική διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως είπα θα ακούμε έναν Ευρωβουλευτή, έναν Εθνικό Βουλευτή. Τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Στέτινα Ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, θα ήθελα να ε, χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία της ε, παρουσίας των βουλευτών από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να επιστήσω την προσοχή στο εξής. Στη Σλοβακία, στην καρδιά της Ευρώπης, εξελέγει πρόεδρος με μεγάλη πλειοψηφία και στην τσεχική δημοκρατία, στη Σλοβακία και ούτω καθεξής γίνονται πολλές ανακοινώσεις σε σχέση με την εκλογή προέδρου, γυναίκας προέδρου στη δημοκρατία τους, της Σλοβακίας λέγοντας ότι θα είναι η αρχή του τέλους για την ομάδα του Βίσενγκραντ. Τι σκέφτεται η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία για την ομάδα του Βίσενγκραντ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σίντε από την Αυστρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εύχομαι καλημέρα σε όλες και όλους για την εξωτερική πολιτική, που είναι το θέμα. Ορίστε, εδώ είμαι, εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, ως πρώτο θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι σημαντικό ε, να υπάρχει μια γνήσια εξωτερική πολιτική της Ένωσης και η αμυντική πολιτική να αποτελεί τμήμα αυτής. Συχνά συμβαίνει το αντίθετο, κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ως σοβαρό σφάλμα. Δεύτερο, μου φαίνεται πραγματικά λυπηρό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν επιτυχάνει συχνά να εμφανίζεται με μια ενιαία φωνή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή στο Δικαστήριο, στο, στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών ή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι σημαντικά τα πράγματα αυτά και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη εάν ενδεχομένω θα πρέπει να κρίνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία. Όταν βλέπω μάλιστα ότι και στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να βρίσκονται αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Σίντερ. Ακολουθεί ο κύριος Αουστρεβίτσιους. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρατε ότι είναι η τελευταία συνάντησή της ΑΦΕΤ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα εξ ονόματος των φιλελευθέρων να εκφράσω την εκτίμησή μας για όλες, όλη την, την όλη συνεισφορά του πρώην Προέδρου, του Έλμαρ Μπρόκ, ο οποίος ε, προώθησε τα θέματα μας μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και παγκοσμίων ε, δεδομένων και εσένα, David. Σε ευχαριστούμε πολύ που προάσπισες ε, τα... που προασπίστηκες των συμφερόντων μας με τόσο καλό και εύγολο το τρόπο. Φυσικά έχουμε να κάνουμε με θεσμικά πλαίσια που θα πρέπει να λειτουργήσουν σωστά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από αυτά τα θεσμικά όργανα. Έχω μία ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την χρονική περίοδο, από το 14 μέχρι το 19, πώς εξελίχθηκε η σχέση μας με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Και θα ήθελα να υποβάλω συγκεκριμένα ερωτήματα πολλές φορές ε, δεν προσδίδουμε τη σωστή σημασία σε ευρωπαϊκά τεκτενόμενα γιατί λαμβάνουν χώρα παράλληλα. Πολλές φορές δίνουμε σημασία, υπέρμετρη σημασία σε ορισμένες περιφέρειες και λιγότερο σε άλλες. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της σκέψης μας και ως προς την όλη μας συνεργασία, πώς κρίνεται αυτή τη συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το επόμενο στάδιο συνεργασίας. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρας, από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ζόλτα Νέμετ από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ, ε, David. Είμαι στον αριθμό 155 εδώ στα έδρανα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που μας κάλεσες και πάλι και ελπίζω ότι αυτός ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και της ΑΦΕΤ θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Όπως άρχισε με τον προκάτοχό σας, τον Έλμαρ Μπροκ και συνεχίζεται και τώρα. Σε σχέση με το έγγραφο, το υποσυζήτηση έγγραφο, νομίζω ότι θα πρέπει να φυγεί το ερώτημα πώς η ΚΕΠΑ μπορεί να γίνει πιο ορατή και πιο αποτελεσματική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε και ιδιαίτερα υπερήφανοι ως προς το μέχρι τώρα έργο μας. Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούσε τα γεγονότα και δυστυχώς ε, οπισθοδρομήσαμε, δηλαδή μπήκαμε σε μία φάση ενδοσκόπησης, ενώ θα έπρεπε να δείξουμε την ηγετική μας θέση. Δεν ήταν δυνατόν όμως να γίνει κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ενδοσκόπηση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τα προβλήματα που μας απασχολούν ιδιαίτερα στην άμεση γειτονία μας. Ας δούμε τι γίνεται με τα Δυτικά Βαλκάνια ή τις σχέσεις μας προς Ανατολάς. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι πολλοί από εμάς ανησυχούμε για τις προκλήσεις την τελευταία διετία. Καλωσορίζω αυτό το έγγραφο. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι και να βρούμε άλλους τρόπους συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Και θα ήθελα να μου πείτε τι, σκέφτεστε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Τι χαρακτήρα θα μπορούσε να έχει. Ως προς την ειδική πλειοψηφία, η άποψή μου είναι αρνητική. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές εξ ονόματος της Ουγγαρίας ότι με βάση την πείρα μας ε, η ειδική πλειοψηφία είναι καθαρά αρνητική όταν είχαμε ειδική πλειοψηφία σε σχέση με την ποσόστοση ε, επανεγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το, η όλη έκβαση αρνητική και ήταν αρνητική επειδή ελήφθη με ειδική πλειοψηφία. Καθώς, και στην ΚΕΠΑ έχουμε τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων με ειδική πλειοψηφία είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το σύστημα. Για παράδειγμα, ένας Έλληνας υπουργός, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά, διορίστηκε ειδικό εκπρόσωπος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ασκήσει το δικαίωμα κυρίας. Νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν είμαστε έτοιμοι. Εάν έχουμε η ειδική πλειοψηφία θα συνεχιστούν οι διχασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε αρκετούς διχασμούς. Θέλουμε να διευρυνθεί αυτό το πλαίσιο διχασμού εισαγάγοντας την ειδική πλειοψηφία. Η θέση μας λοιπόν είναι αρνητική. Θα πρέπει να φτάσουμε σε συμβιβασμούς ο συμβιβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν αναγνωρίσουμε αυτές τις προκλήσεις ενώπιόν μας, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμβιβασμούς, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη θέση της μειοψηφίας, διότι θα οδηγήσει σε μεγάλη διχογνωμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς το έγγραφο, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή μία αρνητική προσέγγιση σε σχέση ε, με το ΝΑΤΟ και τη σχέση μας με την ΙΠΑ, ως προς την Ιερουσαλήμ για παράδειγμα. Γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να επικρίνουμε συνεχώς της ΙΠΑ. Είναι συνετό κάτι τέτοιο. Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε για την πρωτεύουσα του Ισραήλ. Δεν είναι θέμα αυτό εθνικής μάλλον κυριαρχίας και όχι δικό μας. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο αρνητικοί. Εμείς θα πρέπει να χτίζουμε γέφυρες με τις ΙΠΑ και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο. Τέλος, Δυτικά Βαλκάνια. Δεν υποτιμούμε τις απειλές στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία θα πρέπει να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση θα πρέπει να είναι θετική. Κύριε Νέμετ, ε, ήμουνα πολύ γενναιόδωρος και δεν ε, θα μπορούσα να σας δώσω περισσότερο χρόνο δεν βλέπω πρόβλημα, κανένα πρόβλημα με τις εκλογές στη Σλοβακία, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ο Τσάρλς Τάνοκ έχει το λόγο. Δεν θα έπρεπε να είμαι σήμερα εδώ. Ε, είμαστε, θα έπρεπε να ήμασταν στο Brexit συν τέσσερις ημέρες. Είναι βεβαίως πολύ δύσκολη η θέση μέσα στα πλαίσια του κόσμα, του κόμματός μου, με συγχωρείτε του κόμματος των συντηρητικών και δυστυχώς ε, το Κοινοβούλιο ανέλαβε τις ε, διαπραγματεύσεις. Ε, δυστυχώς όμως ούτε χτες έφτασαν σε μια συμφωνία με στα πλαίσια των τεσσάρων επιλογών και νομίζω ότι το ήπιο Brexit δεν πέρασε, μάλλον απορρίφθηκε κατά τρεις ψήφους και η δυνατότητα ε, δεύτερης ενός άλλου ρεφερέντουμ απορρίφθηκε κατά τέσσερις ψήφους. Έχουμε δέκα ημέρες ενώπιον μας πριν από το προσδοκόμενο Brexit και δεν υπάρχει συμφωνία. Ελπίζω να υπάρξει η δυνατότητα ενός δεύτερου δημοψηφίσματος και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι το εκλογικό σώμα έχει αλλάξει θέση, δηλαδή οι νεότεροι ψηφοφόροι θα ψήφιζαν Remain αλλά εν πάση περιπτώσει οι όλες διαπραγματεύσεις είναι ένα είδος εμβολιασμού έτσι ώστε άλλες χώρες να μην αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν οι εθνικοί βουλευτές να συμφωνούν με τον κύριο Τούσκ που βλέπει την μεγαλύτερη εικόνα παραμονής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τελευταία δυόμιση χρόνια προσπάθησα το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν γίνει Brexit, να παραμείνει πολύ κοντά στην ΚΕΠΑ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας είναι πολύ σημαντικό όπου θα πρέπει να συμμετάσχει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είδαμε βεβαίως όμως ότι στο Λονδίνο από όπου προέρχομαι η επιχείρηση ε, Αταλάντα απομακρύνθηκε και θα μεταβεί στην Ισπανία. Όμως το Ηνωμένο Βασίλειο ε, με βάση το γεγονός ότι είναι πυρηνική δύναμη και με όλες μας τις δυνάμεις, τις ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει να μείνουμε κοντά στην ΚΕΠΑ. Δεν θέλουμε να μην υπάρξει συμφωνία και να είμαστε στο χείλος του γκρεμού με βάση την εξωτερική πολιτική ασφαλείας αλλά και την εσωτερική έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την διεθνή τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει όμως να παραμείνουμε κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καλύτερο θα ήταν να παραμείνουμε μέλη. Υπάρχει ε, ακόμα και αυτή την τελευταία στιγμή η δυνατότητα να παραμείνουμε. Ευχαριστούμε. Charles Τάνοκ, υπάρχουν πολλοί ομιλητές, θα ήθελα να αρκεστείτε στα δυόμιση λεπτά. Ο κύριος ε, Μίλο Κόβατς από την Κροατία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ. Θα είμαι πολύ συνεκτικός γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Έτσι θέλω να με θεωρείτε τουλάχιστον. Καταρχήν, δεν νομίζω ότι θα αποδυναμωθεί το ΝΑΤΟ ή θα αποδομηθεί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μπάση περιπτώσει επίσης εμείς θα πρέπει να μιλάμε θετικά ως προς τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Έχουμε έναν ισχυρό δεσμό γιατί εμείς ε, είμαστε η πολιτική δύναμη προς ε, και θα πρέπει να βασιστούμε και στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παραμείνουμε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Τώρα, σε σχέση με την Ήπειρό μας χρειαζόμαστε πράξεις. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με θέματα σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Βλέπουμε όμως μια μεγάλη κρίση στην Ήπειρό μας και βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ είναι ο παράγων που αναλαμβάνει τη σταθερότητα. Δείτε τα Δυτικά Βαλκάνια, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία. Εμείς θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε να ασχοληθούμε με την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβουμε την σταθερότητα της υπήρου μας και να σταματήσουμε να παραπονούμαστε για άλλες χώρες που είναι πιο παρούσες από ό,τι θα έπρεπε. Ευχαριστώ, Μύρο. Ακολουθεί τώρα η κυρία Αλιό Μαρή και επιτέλους αποκαθίσταται λίγο και η ισορροπία μεταξύ των φίλων. Σας ευχαριστώ, David. Τρία σύντομα σχόλια μετά τα όσα άκουσα από ορισμένου εκ των συναδέλφων μας από διάφορες ε, εθνικές βουλές. Πρώτα, η σχέση μεταξύ πολιτικής αμήνης και εξωτερικής πολιτικής. Άκουσα ότι η πολιτική αμήνης υποτάσσεται στην εξωτερική πολιτική. Ως πρώην υπουργό και εξωτερικών αλλά και αμήνης, αυτό αληθεύει σε κάθε χώρα. Στο επίπεδο της Ευρώπης, ωστόσο, είναι διαφορετικά τα πράγματα, διότι δεν έχουμε πραγματική ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, οφείλει να το ομολογήσει κανείς αυτό. Εκτός από θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου είμαστε ενωμένοι, έχουμε πολλές διαφορές και πολλές εντάσεις μεταξύ μας και μόνο με παρεμβάσεων που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε στέλνοντας τους ανθρώπους μας να πάνε να σκοτωθούν στο εξωτερικό, μόνο έτσι ορίζουμε τα πράγματα εκείνα στα οποία συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Δεύτερο σχόλιο για την σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Άμυνας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και ιδίω από την πλευρά τη Ευρώπη. Υπάρχει πραγματική συμπληρωματικότητα. Το ΝΑΤΟ είναι ένα μεγάλο μηχανισμό, πολύ ισχυρό, αλλά και αργό η ευρωπαϊκή άμυνα είναι πολύ πιο ελαφρά αλλά και πολύ ταχύτερη και πολύ πιο εγγύς σε ορισμένες χώρες όπου βλέπουμε πολλαπλές κρίσεις και ιδίως σε χώρες της Αφρικής. Θα πρέπει λοιπόν στην πραγματικότητα να έχουμε μια πραγματική συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο πόλων, όπου η ευρωπαϊκή άμυνα θα επιτρέπει να δρά κανείς γρήγορα, προλαμβάνοντας και κάποιες κρίσεις και εφόσον εξελιχθούν οι κρίσει, τότε βέβαια θα έχουμε ανάγκη από την παρέμβαση του ΝΑΤΟ. Είναι επίση αληθέ ότι υπάρχει και ζήτημα ηγεσία, leadership. Σήμερα οι Αμερικανοί που πάντοτε θέλαν να επιβάλλουν τη δική του ηγεσία, ταυτόχρονα ζητώντα από την Ευρώπη να κάνει όλο και μεγαλύτερε προσπάθειε. Μη λησμονούμε ότι είναι πολύ μεγάλο αισιόδη συνεισφορεύς η Ευρώπη στο ΝΑΤΟ. Ορισμένε ευρωπαϊκέ χώρε, μεταξύ αυτών και η Μεγάλη Βρετανία, την οποία ακούσαμε μόλι πριν, που κάνουν πραγματική προσπάθεια στην άμυνα. Θέλω να πω λοιπόν στους συναδέλφους μου των Εθνικών Βουλών το εξή. Να έχετε συνείδηση ότι σήμερα στην Ευρώπη η προσπάθεια άμυνας και ασφάλειας που κάνουν οι πολίτες, δηλαδή με τους φόρους που καταβάλουν, είναι, η διαφορά είναι από 1 έως το 10. Βλέπει Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία που κάνουν μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή ε, δαπάνες και άλλε που δεν κάνουν τίποτε, επειδή βασίζονται στις πρώτες. Όμω η κατάσταση παγκοσμίω είναι πολύ επικίνδυνη. Ποτέ δεν ήταν τόσο επικίνδυνη και θα γίνεται όλο και περισσότερο. Και λόγω κρίσεων σε τρόφιμα, περιβάλλον κλπ. Ο καθένα λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε του και κάθε Εθνική Βουλή θα πρέπει να δεχθεί να αυξήσει τον αμυντικό προπολογισμό τη. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Αριομαρή. Η ε, κυρία Ντεριδά από την Γερμανία ε, βουλευτή τη Γερμανική Βουλή. Ευχαριστώ. Μπορώ να ε, συνδέσω την ομιλία μου ακριβώ με αυτό που είπε η κυρία Λιωμαρή. Είναι πράγματι σημαντικό και σωστό να έχουμε κοινή εξωτερική στρατηγική. Όχι μόνο για τα όσα λέχθηκαν ω τώρα σε ό,τι αφορά την Ατλαντική Συμμαχία. Όποιος πίστεψε στην αρχή ότι θα ξεφορτωθούμε γρήγορα τον πρόεδρο Τραμπ θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη και την γνωμοδότηση που εξέδωσε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008 και που λέει καθαρά πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχή. Χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια και για τις επιμέρους χώρες και τις κυρίαρχες στρατηγικές τους. Και όταν μιλούμε για ένα ταμείο, δεν θα πρέπει να μιλήσουμε μονάχα για αμυντικό ταμείο το οποίο θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση των εξοπλιστικών βιομηχανιών που κάνουν εξαγωγέ. Πρέπει να μιλήσουμε για ένα ταμείο συνοχή και αυτό να τροφοδοτείται χρηματοδοτικά. Όχι, δεν είμαστε υπέρ τη αποβιομηχάνηση. Και γι' αυτό πρέπει να σκεφτείτε καλά και την οδηγία για τι εξαγωγέ εξοπλισμών. Και εδώ χρειάζεται ευρωπαϊκή οδηγία η οποία να έχει ισχυρό δεσμευτικό χαρακτήρα. Να επανέλθω όμως στην έκθεση. Η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας μου φαίνεται εξαιρετική. Τονίζω όμως ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη πολύ περισσότερο τις γυναίκες και την ειρήνη. Πολύ περισσότερο από ό,τι το πράττει στην παράγραφο 20. Γνωρίζουμε ότι όταν οι γυναίκες συμμετέχουν στις ειρηνευτικές διαδικασίες, αυτές είναι πολύ πιο αποτελεσματικές. Και γι' αυτό θέλω να ενισχυθεί πολύ το κείμενο της παράγραφου αυτής. Και τέλος, για την διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση. Εδώ τίθεται το ερώτημα πώς θα ε, τονίσουμε περισσότερο την ψηφιοποίηση της αμυντικής πολιτικής. Γνωρίζουμε ότι αναπτύσσονται συστήματα και εδώ πρέπει να δούμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα πολύ εντονότερα από ό,τι έχουμε πράξει έως τώρα. Και εδώ επανέρχομαι στο θέμα της ισότητας των φύλων, αλλά όχι μόνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μην έχουμε ένα σύνολο κανόνων όπως έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Για να ενισχυθεί και η εσωτερική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως χωρίς στρατηγικές εξυγχρονισμού αυτά τα βήματα δεν θα επιτύχουν. Ευχαριστώ κυρία ε, Ρίντερ θα ακολουθήσει ο ευρωβουλευτής του EFTD, James Carver, επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μου φαίνεται ότι μάλλον όμως αυτός θα είναι υπέρ του Brexit. David, ε, ε κατά πάθα η τελευταία μου παρέμβαση ως Βρετανού Ευρωβουλευτού και θα ήθελα να απευθύνω φόρο τιμής σε εσά, κύριε Πρόεδρε, διότι Είστε απολύτως αντίθετος πολιτικά από εμένα, αλλά φροντίσατε πάντοτε να ακούγεται η γνώμη μου. Και σας ευχαριστώ. Πάντοτε υπήρξατε απολύτως έντιμος και αντικειμενικός. Έτσι θα πρέπει να εργάζεται κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω για το Brexit, δεν είναι ο κατάλληλος τόπος. Αυτά που συζητούμε εδώ τώρα είναι αμυντική πολιτική και εξωτερική πολιτική. Ε, Ιδίω δηλαδή η δική πλειοψηφία. Ακούσαμε σήμερα το πρωί συχνά περιπεπρωμένου σε σχέση με τις εξωτερικές υποθέσεις. Δεν νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές μπορούν να δώσουν εντολή για τέτοια πράγματα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και πολύ σοβαρό. Και θα επηρεάσουν το μέλλον των 27 χωρών μελών πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε χώρες όπως Αυστρία και Σουηδία που είναι παραδοσιακά αδέσμευτες. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή για το τι θέλετε. Από συζητήσεις που έχω διεξαγαγεί και η γυναίκα μου μάλιστα είναι Νορβηγίδα, χρειάζεται να προσέξετε πάρα πολύ διότι θα μπορεί να ε, οδηγήσουν σε επιζήμιες συνέπειες τέτοιες συζητήσεις. Μην προσπαθείτε να διορθώσετε κάτι που λειτουργεί. Το ΝΑΤΟ έχει λειτουργήσει θαυμάσια όλα αυτά τα χρόνια και το λέω σε εσά του εκπροσώπου τη Ευρώπη των 27, αναρωτηθείτε στα σοβαρά τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να υλοποιήσει το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ κύριε Κάρβερ. Ακολουθεί ο κύριος Ρόχας από την Ισπανία. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μακάλιστερ για την πρόσκληση. Μιλάμε για τη μετανάστευση. Το θέμα της μετανάστευσης είναι μία από τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα, γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο μέλλον με βάση την αλληλεγγύη και την αμοιβαία ευθύνη θα πρέπει να έχουμε βεβαίως έλεγχο των συνόρων, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τις διάφορες μαφίες που δρούν στα σύνορα. Θα πρέπει να δούμε ποιοι ευεργετούνται από αυτή την παράνομη μετανάστευση και να τους αντιμετωπίσουμε. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις συνιστώσεις του προβλήματος και ένας προγραμματισμός από τους Ευρωπαίους εταίρους. Έτσι θα έχουμε μια τακτική και σίγουρη μετανάστευση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις διάφορες μαφίες. Αυτός είναι ένας τους πυλώνες συνεργασίας κατά της ε, παράνομης μετανάστευσης. Θα πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη με το ΝΑΤΟ και τις γειτονικές ε, ε, χώρες, διότι υπάρχει ένας τζίρος 700 δις και στην ουσία πρόκειται για μια κατάσταση σκλαβιάς εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει διάφορα μέτρα για να σταματήσει αυτή η διακίνηση που γίνεται από τις διάφορες μαφίες. Χρειάζεται όμως συνεργασία Frontex και άλλων οργανισμών μέσα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ όπως το Τρίτον Ποσειδών ή την επιχείρηση Σοφία οι επιχειρήσεις είναι επιτυχείς καταρχήν, αλλά κατανοούμε ότι δεν επαρκούν, γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε αυτή την σημαντική αποστολή. Ευχαριστώ. Ακατόπιν, ο κύριος Ιβο Βάγγελ, Ευρωβουλευτής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη Σλοβενία είμαι και βλέπω πως υπάρχει και μια μικρή αντιπροσωπεία από την Βουλή της Σλοβενίας. Θα προσπαθήσω να τους κάνω αισθανθούν πιο άνετα, να μιλήσω τη γλώσσα μας. Είμαι ευρωβουλευτής ε, εδώ και 10 χρόνια, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών. Τώρα που φεύγω από αυτό το κοινοβουλίο αισθάνομαι μια θλίψη. Θεωρώ ότι ο κόσμος τώρα είναι πολύ πιο επικίνδυνος από ότι ήταν πριν από 10 χρόνια όταν έγινε ευρωβουλευτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έγινε παγκόσμιος παίκτης, δεν κάθεται ε, στα τραπέζια που λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, περί ειρήνης ή πολέμου. Και βεβαίως τα θέματα ειρήνης και ασφαλείας είναι η ουσία της ε, πολιτικής άμυνας και ασφαλείας. Γι' αυτό έχουμε ένα μέσο που λέγεται διεθνές δίκαιο στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Δυστυχώς ε, δεν το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά. θεωρώ ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε την σημασία του διεθνούς δικαίου στα πολυμερή φόρουμ, στο διμερές πλαίσιο και στην επίλυση των προβλημάτων. Μόνο εάν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο και το θεωρούμε βάση για την επίλυση διεθνών προβλημάτων, θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για προβλήματα όπως το μεσανατολικό, το πρόβλημα της Δυτικής ε, Σαχάρας, ε, Ουκρανίας και τα λοιπά τώρα μπορώ να σας πω πολλά. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Ε, δεν θεωρώ ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις με την δημιουργία πλειοψηφιών όταν λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται μια ισχυρή ηγεσία η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητάμε πολύ περισσότερο. Μόνο έτσι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει σημαντικός παίκτη στην διεθνή σκηνή. Σας ευχαριστώ. Κατόπιν έχουμε τον κύριο Μπιζέ από την Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μακάλιστερ θα ήθελα καταρχήν να πω ότι με αυτά που είπε η συνάδελφος Μισελ Αλιομαρή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ που αποτελούν συμπλήρωμα ο ένας φορέας του άλλου. Σε σχέση με τη δημοσιονομική προσπάθεια η Πολωνία το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες προς την προσπάθεια αυτή. ή θα ήθελα να συμμετάσχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο στο ΝΑΤΟ, να συνεισφέρουμε περισσότερο. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε, διότι προσδίδοντας μεγαλύτερη σημασία και δίνοντας περισσότερα χρήματα στο ΝΑΤΟ, όπως κατανόησαν οι Αμερικανοί εδώ και δεκαετίες, μπορούμε να επηρεάσουμε τα ε, πράγματα περισσότερο. Τώρα, ως προς το πέρασμα στην ειδική πλειοψηφία, νομίζω ότι είναι απολύτως αναγκαίο, γιατί όταν υπάρχει μόνο ομοφωνία υπάρχει και παράλυση εργασιών. Θα πρέπει κανείς να μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα καλύτερα. Νομίζω λοιπόν ότι μία στάθμιση ψήφων είναι το καλύτερο σύστημα. Εάν στην, σε θέματα ΚΕΠΑ δεν περάσουμε στην ειδική πλειοψηφία, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληγεί ιδιαίτερα, θα παραλύσει. Και τα οικονομικά και ε, στρατιωτικά δρόμενα κινούνται πολύ πιο γρήγορα από την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Άρα, εάν δράσουμε ομόφωνα, τότε θα επιβραδύνουμε τις όλες διαδικασίες. Στην προσεχή θητεία, λοιπόν, θα πρέπει να περάσουμε στην ειδική πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Κατόπιν, ο κύριος Κρίστιαν Πρέντα, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Δύο λόγια επιτρέψτε μου πρώτα να πω για την ε, ειδική πλειοψηφία. Είμαι απολύτως υπέρ, διότι θεωρώ μετά από δεκαετή συμμετοχή μου εδώ και τα πέντε μάλιστα χρόνια ως συντονιστής, βλέπω επί του πεδίου πώς οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς εργάζονται και οι αντιπροσωπείες των χώρων μελών και διαπιστώνω ξανά και ξανά ότι η αδυναμία της Ευρώπης συνίσταται πράγματι στην αρχή του συμβασμού που έχει, την έχει κάνει απόλυτο κανόνα και της ομοφωνίας εννοείται. Επιτρέπει έτσι και ας πούμε ανέντιμες συμμαχίες οι οποίες μπλοκάρουν ξεκάθαρες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα των ε, εξωτερικών σχέσεων. Δεύτερο, βρίσκω επίση σημαντικό το φάκελο των Δυτικών Βαλκανίων και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και ο επόμενος επίτροπος αρμόδιος για τη διεύρυνση, εφόσον υπάρχει τέτοιο χαρτοφυλάκιο, θα πρέπει να ρίξουν το βάρος τους στην διεύρυνση. Ο ρυθμός και η μεθοδολογία πάσχουν και υπάρχει κίνδυνος να τα χάσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να γίνει πολιτική προτεραιότητα, γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία για εμάς τους Ευρωπαίους. Σας ευχαριστώ. Thank you, Christian Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους τέσσερις τελευταίους ομιλητές. Ε, ο κύριος Μπένσεκ από την Τσεχία, ο κύριος Καμεντσίνη από την Ιταλία, η κυρία Μάνταλα από τη Γερμανία και ο κύριος Βοσκεβιτς από την Πολωνία. Ξέχασα κάποιον? Όχι. Αυτοί είναι οι τέσσερις τελευταίοι ομιλητές. Ο κύριος Μπένετσακ πρώτος. Ο κύριος Στέτινα μας ε, πρότεινε να μιλήσουμε για την ομάδα του Βίσεγκραντ. Εγώ ως ε, πρόεδρος της ε, Βουλής των Κοινοτήτων υπεύθυνο για ευρωπαϊκά ζητήματα μπορώ να σας πω ότι διαθέτουμε μία επίσημη πλατφόρμα γίνονται συναντήσεις δύο φορές το χρόνο και μπορώ να σας πω ότι τα θέματα που μας απασχολούν επιλέγονται κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ουσιαστική και διασταυρούμενη συζήτηση. Ε, δεν ε, είμαστε μία μονολυθική οντότητα όπως μας παρουσιάζουν πολλοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ούτε είμαστε ταραχοποιοί. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό. Και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν πολλές αποχρώσεις γιατί η Πολωνία ψήφισε υπέρ των ποσοστώσεων, ενώ η Τσεχία δέχτηκε να υποδεχτεί περισσότερους μετανάστες σε εθελούσια βάση, άρα κανένας δεν επιβάλλει κάτι. Η Ουγγαρία ένα χρόνο μετά δέχτηκε χίλιους μετανάστες και η Σλοβακία το 1% για να τηρήσει την ποσόστοση. Μετά ο πρόεδρος μας έλαβε το λόγο και είπε ότι η ομάδα του Βίσεγκραντ έπεισε τους πάντες ότι η κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει. Κατανοώ ότι πολλοί συνάδελφοι βλέπουν την ομάδα του Βίσεγκραντ υπό αυτό το πρίσμα, αλλά όσον αφορά το μέλλον όλα εξαρτώνται από εμάς κατά μείζωνα λόγο και αυτές οι περιφερειακές οντότητες ε, δεν αποτελούν εξαίρεση στην Ευρώπη. Θα μπορούσα να μιλήσω για το Μπενελούξ. Σε σχέση με αυτά που προελέχθησαν, νομίζω ότι χρειάζεται μία συμπληρωματική πολιτική σε σχέση με αυτή του ΝΑΤΟ. Γιατί γιορτάζουμε 25 χρόνια μετά την προσχώρησή μας στο ΝΑΤΟ και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι διακοινοβουλευτικές συζητήσεις ως προς την εξωτερική πολιτική ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Χαίρομαι λοιπόν γιατί έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την έκθεση, αλλά θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσέξει ιδιαίτερα ως προς τις επιλογές του. Thank ευχαριστώ. Ε, ίσως είδατε τις κάμερες πριν συνεχίσουμε να καλωσορίσω τον ε, κύριο Μπαρνιέ στη συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε. Έχετε, έχετε πέντε λεπτά ακόμα να περιμένετε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κομεντσίνη λοιπόν από την Ιταλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να λάβω θέση επί δύο ζητημάτων. Να μιλήσω για τον αντιφατικό χαρακτήρα αυτής της πρότασης, να περάσουμε δηλαδή από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία, Σημερίζουμε τη γνώμη πολλών συναδέλφων ότι δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο στρέφεται κατά της εθνικής κυριαρχίας και τις διάφορες ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες που ενυπάρχουν στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και θα θέλαμε να εκφράσουμε αρνητική γνώμη. Ως προς το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, συμμερίζομαι αυτά που είπε ο Ισπανός συνάδελφος υπό την έννοια ότι πολλές μελέτες έδειξαν ότι η Ιταλία και η Ισπανία βρίσκονται μόνες τους και πρέπει από μόνες τους να αντιμετωπίσουν αυτό το μείζον πρόβλημα. Επίσης, πολλές φορές ε, υπάρχει πίσω από όλα αυτά το οργανωμένο έγκλημα το οποίο διακινεί ανθρώπους και κερδοσκοπεί δυστυχώς εις βάρος αυτών των ανθρώπων έχοντας πολύ υψηλά έσοδα. Θα πρέπει λοιπόν να αναχαιτιστεί αυτή η πορεία και η Ευρώπη να παίξει το δικό της ρόλο. Η Frontex από ό,τι μάθαμε χτες θα ενισχυθεί αλλά περιμένουμε συγκεκριμένες εξελίξεις, διότι η Ιταλία όπως και η Ισπανία και η Ελλάδα είναι μόνες τους στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Και αυτό πέρα από, την οργανωμένη, από το οργανωμένο έγκλημα δείχνει ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος στην Ευρώπη από την παράνομη μετανάστευση γιατί πολλοί τζιχαντιστές ή άλλα εγκληματικά στοιχεία, τρομοκρατικά στοιχεία θα μπορούσαν να μεταβούν στην Ευρώπη. Θεωρούμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό γιατί καταρχήν θα πρέπει να μπορούν να ε, εγκατασταθούν και να επαναπατριστούν στην χώρα τους. Κυρία Μάνταλα από Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λόγω του προκεχωρημένου της ώρας έχω μόνο ένα μήνυμα να σας μεταφέρω από την Γερμανία. Εμείς είμαστε αξιόπιστος εταίρο του ΝΑΤΟ και θα είμαστε μόνο εφόσον λειτουργούμε συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ τη ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης, εφόσον την επεξεργαζόμαστε και αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο. Για αυτό το λόγο το κοινό Συμβούλιο Άμυνα είναι σωστό, σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τις αιτίες για την ε, εγκατάλειψη των αισθειών των ανθρώπων και πρέπει να εμφανιστούμε ως αξιόπιστοι εταίροι του ΝΑΤΟ καταπολεμώντας από κοινού την τρομοκρατία και να συνεχίσουμε να φροντίζουμε ώστε και άλλες χώρες να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ευχαριστώ ρητά τον κύριο Τάνοκ για την σημερινή του παρουσία εδώ, τον Βρετανό Ευρωβουλευτή που μίλησε προηγουμένως. Και είναι ένα σημάδι αυτά που είπε πόσο, για το πόσο σημαντική είναι η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Τελευταίος ο κύριος Βοσικίβιτς από την Πολωνία. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να είμαι σύντομος. Η σημερινή συζήτηση ε, βρίσκω ότι έχει εξαιρετική σημασία. Πολλοί από αυτούς ε, που προηγήθηκαν εμού στο μικρόφωνο τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η ειδική πλειοψηφία αλλά και η ομοφωνία. Όμως θα πρέπει να είναι κατανοητές οι απόψεις όλων των χωρών μελών. Γιατί αλλιώς δεν θα, έχουμε, δεν μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή ενότητα, ιδίως για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ο συνάδελφος μας από τη Σλοβενία ρώτησε πώς βλέπουμε την ομάδα Βίσεγκραντ. Εμείς θεωρούμε όλοι ότι πρέπει να συνομιλούμε μεταξύ μας. Το θέμα της ε, ειδικής πλειοψηφία έχει ιδιαίτερη σημασία. Όμως πώς θα διαμορφωθεί αυτή η ειδική πλειοψηφία. Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε και να το αποφασίσουμε εμείς σήμερα εδώ. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να προσεγγίζει την απόλυτη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ όλες και όλους για τις παρεμβάσεις σας, μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέρουσες ε, και καλύψατε όλο το φάσμα των ε, διαφόρων ε, απόψεων για την ε, λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στην εξωτερική πολιτική. Το ίδιο Μιλήσατε και τοποθετηθήκατε και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλεία. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και είμαι βέβαιο ότι στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο θα αποτελέσουν σημαντικά θέματα γύρω από τα οποία θα στραφεί η συζήτηση που θα διεξαχθεί και στην παρούσα Επιτροπή. Γιατί και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών μα αναμένει από εμά να προχωρήσουμε. Βεβαίω, συχνά, όπω λένε και οι Αγγλοσάξονε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας. Εν τω μεταξύ θα ήθελα βέβαια να προχωρήσουμε στο θέμα υπαριθμών 10 της ε, κανονικής μας ημερήσιας διάταξης με πρώτο σημαντικό θέμα την κοινή συνεδρίαση ε, και πάλι σας καλωσορίζω κύριε Μπαρνιέ σήμερα στην κοινή συνεδρίαση των μελών Τη επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ομολόγων μας εθνικών βουλευτών των αρμόδιων, συναρμόδιων μάλλον επιτροπών. Λίγα λόγια πρώτα για το Κοινοβούλιο. Εγώ είχα την εντύπωση ότι τους τελευταίους μήνες, για να μην πω χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε να μεταφέρει τις θέσεις μας στην Brexit Steering Group και ταχθήκαμε πάντοτε υπέρ των προσπαθειών των συντονιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπάθειες που ήταν ουσιώδεις έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλεί με μια φωνή. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Μισελ Μπαρνιέ και σε ολόκληρη την ομάδα του για την σκληρή δουλειά που έκαναν τα τελευταία αυτά χρόνια υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενότητα των χωρών μελών της. Η διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Αποχώρησης και η πολιτική δήλωση δεν ήταν βέβαια απλά πράγματα. Υπήρξαν πολύ, αποτέλεσμα πολύ, σκληρή, πολύ σκληρής και σε αχαρτογράφητα ύδατα. Ορισμένες από τις πτυχές της ε, Συμφωνίας Αποχώρησης αναφέρονται και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όπως και ΠΑ και πολιτική ασφάλειας Είμαι βέβαιος ότι θα μα ε, μιλήσει για τα πράγματα αυτά ο Μισελ Μπαρνιέ. Σα ευχαριστώ και πάλι που είστε σήμερα εδώ. Γνωρίζουμε πόσο πολύ άσχολο είστε και ιδίω μετά από τα χθεσινοβραδινά ε, γεγονότα στην Βουλή των Κοινοτήτων ε, τη μεγάλη Βρετανία. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Θα ακούσουμε τι αγωγικέ σα παρατηρήσει και μετά έχουμε χρόνο με περίπου μία ώρα για ερωτήσει και απαντήσει. Έχετε το λόγο, Μισελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα σε όλους. Δεν είναι υποχρεωτικό να μιλάω αγγλικά. Ωραία, θα μιλήσω γαλλικά λοιπόν. Ε, απλά για να σας ε, δείξω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτή την ε, ποικιλομορφία. Αγαπητέ Ντέιβιτ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Όπως ξέρετε είμαι πολιτικός και στην πολιτική μου πορεία γνώρισα στιγμές ή φάσεις που ήταν καθοριστικές. Ήμουνα υπουργό Εξωτερικών, ήμουν διαπραγματευτής διαφόρων συνθήκων, ιδιαίτερα της συνθήκης της Λισαβόνας, σε σχέση με θέματα ευρωπαϊκής άμυνας. Άρα καταλαβαίνετε ότι με απασχολούν εκ του τα ζητήματα που απασχολούν και εσάς. Τα αντιμετωπίζω με δυναμισμό όπως και εσείς. Στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων ή στην Επιτροπή Άμυνας. Για 20 χρόνια ήμουν εθνικός βουλευτής, με ευχαριστείτε που βρίσκομαι εδώ, εγώ όμως σας ευχαριστώ, γιατί αυτή η διαπραγμάτευση που ε, διάγω εδώ και δύο χρόνια ε, δεν ε, ήταν εμπιστευτικού χαρακτήρα. Επισκέφτηκα τα 28, 27 μάλλον κοινοβούλια, εθνικά κοινοβούλια και βεβαίως και τους Βρετανούς. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Πολωνία, αύριο θα είμαι στη Σουηδία. Συνεχίζω αυτή την εργασία και σε κάθε επίσκεψη επισκέφτομαι τα εθνικά κοινοβούλια, διότι είναι ένα θέμα που σας αφορά άμεσα. Αυτή η διαπραγμάτευση που αφορά τόσα εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη. Πέρα από αυτό το διαζύγιο λοιπόν που προσπαθούμε να οργανώσουμε, το θέμα μας απασχολεί. Δεν θέλουμε μία άτακτη αποχώρηση. Υπάρχει και μία δεύτερη διαπραγμάτευση που αφορά τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη μελλοντική εταιρική σχέση. Και το σύνολο αυτής της εταιρικής σχέσης, πέρα από την ΚΕΠΑ, αφορά ζητήματα που θα περάσουν σε μικτές συμφωνίες. Δηλαδή, κάθε εθνικό κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί. Τα 27 εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αποφανθούν ομόφωνα για τη μελλοντική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα άμεσα. Θα μεταβώ σε κάθε πρωτεύουσα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, το χρόνο και την υποστήριξή σας, που είναι μια συλλογική υποστήριξη μέσα στα πλαίσια της Σαμπίν Βεγιάν Στεφανή Ριζό, της ομάδας δηλαδή που με πλαισιώνει. Ζούμε δύσκολες στιγμές στη διαπραγμάτευση αυτή. Βρισκόμαστε στον αέρα με βάση τις αποφάσεις του Βρετανικού Κοινοβουλίου ως προς τη ε, συνθήκη που διαπραγματευτήκαμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη συμφωνία αυτή δηλαδή. Εδώ και τέσσερις μήνες υπάρχει αυτή η συμφωνία για την τακτική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 600 σελίδες. Κατανοώ ότι δεν μπορεί κανείς να διαβάσει εύκολα το κείμενο και υπάρχει ένα δεύτερο ε, μέρος του κειμένου. Αυτό το κείμενο το δείχνει ο Μισελ Μπαρνιέ. Το συνοδευτικό κείμενο, δηλαδή της αποχώρησης και όπως ξέρετε σε κάθε διαζύγιο θα πρέπει να αποφανθούμε επί του παρελθόντος, να φτάσουμε σε μία συμφωνία και να ορίσουμε την πορεία για μία μελλοντική, σημαντική εταιρική σχέση με αυτή τη μεγάλη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, μάλλον το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ψήφισε χτες με αρνητική ψήφο για όλες τις εναλλακτικές, αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό, διότι η Βουλή των Κοινοτήτων της χώρας αυτής που αποφάσισε να αποχωρήσει από, το Ηνωμένο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγχωρείτε, δυστυχώς δεν εγγράφεται καμία θετική πλειοψηφία. Υπάρχουν αρνητικές πλειοψηφίες κατά της συμφωνίας, κατά της μη συμφωνίας και κατά όλων των άλλων εναλλακτικών λύσεων. Αν και είναι μικρές αυτές οι αποκλίσεις. Είδατε χτες τι συνέβη σε σχέση με ενδεχόμενη τελωνιακή ένωση. Χάθηκε αυτή η εναλλακτική με δύο ψήφους. Αλλά έτσι δεν μπορούμε να οργανώσουμε την τακτική αποχώρηση του Ηνωμένου ε, Βασιλείου. Για να μην υπάρξει άτακτη αποχώρηση, θα πρέπει κάτι να ψηφιστεί για τακτική αποχώρηση. Εάν λοιπόν υπάρξει τακτική αποχώρηση, υπάρχει μόνο μία ενδυνάμει συμφωνία. Είναι αυτή που βλέπετε. Την διαπραγματευτήκαμε, διαπραγματευτήκαμε όλα τα επιμέρους στοιχεία αυτής της συμφωνίας για να μην για να υπάρχει ακριβώς νομική ασφάλεια και να μην υπάρχει καμία ασυμφωνία. Άρα το no deal, η άτακτη δηλαδή αποχώρηση, ε, διαφαίνεται στον ορίζοντα. Είμαστε προετοιμασμένοι, δεν είναι η δική μου επιλογή, δεν χρειάζεται κανείς διαπραγματευτεί για ένα no deal, αλλά για μια συμφωνία. Είμαστε όμως έτοιμοι εδώ και αρκετούς μήνες για αυτό το ενδεχόμενο. Όπως καταλαβαίνετε το Brexit μονοπόλησε τις συζητήσεις μας το τελευταίο καιρό, δαπανίσαμε πολύ χρόνο και ενέργεια και γι' αυτό τώρα θα πρέπει να βρούμε μια θετική ατζέντα. Θυμάμαι ότι η καγκελάριος η Άγγελα Μέρκελ στην απαρχή της διαδικασίας έλεγε ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό από το Brexit. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τις πραγματικές προκλήσεις που διαγράφονται. Ελπίζω να έχουμε θετική έκβαση της διαπραγμάτευσης και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που είναι ολοένα και πιο σοβαρές, κλιματικές αλλαγές, οι οικονομικές προκλήσεις, ο τεχνολογικός πόλεμος, η μετανάστευση, η ευρωπαϊκή άμυνα και ούτω καθεξής. Ο πρόεδρος Γιούνκερ από την αρχή της θητείας του, εδώ και τέσσερα χρόνια, όρισε μία φιλόδοξη ατζέντα και για την προστασία βεβαίως των επενδύσεων και το μεταναστευτικό. Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Τούσκ πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ασχοληθεί με μείζονο σημασία ζητήματα όπως οι βιομηχανικές εξελίξεις και πολιτική και οι σχέσεις μας με την Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τον κόσμο όπως διαγράφεται, όπως διαμορφώνεται με τη διασπορά των απειλών που διεισδύουν όλο ένα και περισσότερο τον κοινωνικό μας ιστό με την σωστή λειτουργία της, ε, δύο, δημοκρατίας, την τρομοκρατία, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις εξωτερικές επεμβάσεις, καθώς και την αμφισβήτηση ορισμένων θεμελιωδών αρχών της συλλογικής ε, ασφάλειας, τη, τους κλειδονισμούς στο ε, ΝΑΤΟ, την παλινοδία των ΗΠΑ και τις ε, πολυμερείς μας σχέσεις. Και εν γέννη θα πρέπει να μην δεχτούμε τον προστατευτισμό των ΗΠΑ και να δούμε και θέματα ως προς τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και την νέα υπερδύναμη που ανακύπτει, δηλαδή την Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν να μην αποδυναμωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να είναι το κεντρικό μας μέλημα. Αυτό αφορά τις σχέσεις μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν και θέματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα μία συζήτηση με τον Νάιτζελ Φαράζ. Ξέρετε για ποιον ε, μιλάω. Στο τέλος αυτής της συνομιλίας ε, ζήτησα, ρώτησα μάλιστα τον κύριο ε, Φαράζ του εξής. Κύριε Φαράζ, κάνατε μία εκστρατεία υπέρ του Brexit. Κερδίσατε, το σεβόμαστε, λυπούμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συμφωνία για το Brexit. Μπορείτε να μου πείτε όμως πώς βλέπετε τα πράγματα μετά το Brexit. Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι μελλοντικές μας σχέσεις, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μεγάλη Βρετανία. Η απάντησή του ήταν σαφέστατη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξής. Κύριε Μπαρνιέ, μετά το Brexit η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπάρχει πια. Αυτό μου απάντησε. Άρα θέλει, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των έσω. Όπως άλλοι προσπαθούν να το κάνουν από το εξωτερικό, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, πολλές πολιτικές μας πρέπει να τις ε, επανεξετάσουμε ως προς την επικουρικότητα, να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Σίγουρα χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, θα πρέπει να αντλήσουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να υπερασπιστούμε τα γενικά μας συμφέροντα. Προσπάθησα να το κάνω μέσα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης αυτής. Νομίζω ότι η διπλωματία, η άμυνα, η ανάπτυξη, η συνεργασία με άλλες περιφέρειες του κόσμου, καταρχήν με την Αφρική, είναι οι τρεις ε, μεγαλύτεροι μοχλοί για να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκακέρα. Θα πρέπει στο μέλλον να ενισχύσουμε τις διπλωματικές μας ικανότητες για να μιλάμε με μία φωνή, να μην είμαστε διχασμένοι όπως ίσχυσε στην περίπτωση της Βενεζουέλας ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις απειλές χρησιμοποιώντας τις 140 αντιπροσωπείες μας ανά τον κόσμο. Να ενισχύσουμε την ειδική πλειοψηφία Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Επίσης, να προτάξουμε την εξωτερική μας δράση. Εμείς είμαστε ο πρώτος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι με βάση τα δικά μας συμφέροντα, ανησυχίες και προσδοκίες έναντι ορισμένων χωρών και γι' αυτό η διπλωματία μας θα πρέπει να λάβει υπόψη και οικονομικές και εμπορικές συνιστώσεις. Τέλος, θα πρέπει να προωθήσουμε τις προσπάθειες υπέρ της ευρωπαϊκής ασφάλειας, να προστατεύσουμε την ήπειρό μας και βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις η πρώτη προσδοκία των Ευρωπαίων πολιτών, ε, και αυτό δεν είναι παράδοξο, είναι η ΚΕΠΑ το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις εθνικές προσπάθειες που γίνονται και με την κοινή προσπάθεια στα πλαίσια της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και το Ηνωμένο Βασίλειο και τις, τη διμερή συνεργασίες που έχουμε με πολλές χώρες όπως και τη Μεγάλη Βρετανία. Να προστατεύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας παντού ανά τον κόσμο να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις στην πηγή τους και να προγραμματίσουμε καλύτερα το μέλλον. Αυτή η φιλοδοξία που σας κυαγράφησα σχετίζεται με τη συνεργασία των 27. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε μια στενή εταιρική ε, σχέση με, τη Μεγάλη Βρετανία, όπως είπατε και εσείς κυρία Μοντερλά στην παρέμβασή σας. Ε, διπλωματία, συνεργασία, άμυνα, έτσι ώστε να χτίσουμε μία βιώσιμη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η πολιτική δήλωση που σας δείχνω και θα ήθελα να διαβάσετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και προωθούμε με την ομάδα της ε, Τερέζα Μέη. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σύμμαχός μας στα πλαίσια του Μονίμου Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχουμε κοινά συμφέροντα και είμαστε αλληλέγγυοι ως προς τις ενδεχόμενες εξωγενείς απειλές. Και γι' αυτό ακριβώς εδώ και έναν χρόνο, πέρσι τον Ιούλιο, συνεργαστήκαμε και εργαστήκαμε ως προς τα δικά σας ψηφίσματα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τη λευκή βίβλο που προτάθηκε τον Ιούλιο από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κάναμε ένα συγκεκριμένο benchmarking για να βρούμε τα σημεία σύγκλησης. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για όλα αυτά και έχει επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος. Θα ήθελα να μιλήσω για τους πέντε μηχανισμούς που ορίσαμε με το Ηνωμένο Βασίλειο και επί των οποίων θα συνεργαστούμε. Πρώτον, στρατηγικός διάλογος για κοινέ προσπάθειες στα Ηνωμένα Έθνη μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας να απαντήσουμε στις μεγάλες ε, προκλήσεις, δηλαδή διάδοση πυρηνικών από το Ιράν, κλιματικές αλλαγές, καθώς και πολιτικός και στρατηγικός διάλογος για το κυρωτικό πλαίσιο που θα επιβάλλουμε. Δεύτερον, λειτουργική συνεργασία έτσι ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο, αν το επιθυμεί, να συμμετάσχει στη διαδικασία σταθεροποίησης μέσα στα πλαίσια καταπολέμησης της πειρατείας στον κόλπο του Άντεν ή στον Περσικό κόλπο, καθώς ε, και ε, τις στρατιωτικές δυνάμεις που εκπαιδεύονται στη Σομαλία να συνεργαστούν μαζί μας για αυτή την ε, επιχειρησιακή συνεργασία εκτός Ευρώπης. Τρίτον, τη δυνατότητα συμμετοχής σε σχέδια έρευνας και στρατιωτικών επιχειρήσεων για να υπάρχει διαλειτουργικότητα ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και της νέας συνεργασίας, μόνιμης συνεργασίας το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε την, ε, την δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές τις ε, κοινέ προσπάθειες στρατιωτικής συνεργασίας και μόνιμου μηχανισμού. Τέταρτον, ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μη διάδοση πυρηνικών όπλων ή υβριδικών όπλων αντιμετώπιση νέων απειλών μέσα στα πλαίσια του κυβερνοχώρου, της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, μέσα στα πλαίσια των διεθνών συνθήκων και με όλους τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί που αναγνωρίσαμε με τους Βρετανούς και που έχουμε εντάξει σε αυτή την πολιτική δήλωση και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε το ταχύτερο δυνατόν υπό την αίρεση ότι θα υπάρξει συμφωνία για το διαζύγιο και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέραν από αυτά, είχαμε προβλέψει και μία συνεργασία ασφάλειας μέσα στα πλαίσια μεταβατικών μέτρων, έτσι ώστε αυτή η εταιρική σχέση να τεθεί σε εφαρμογή πριν από το τέλος της μεταβατικής φάσης. Μία ευέλικτη εταιρική σχέση χωρίς υπερβολική κωδικοποίηση με βάση τα συγκλίνοντα συμφέροντα και μία εταιρική σχέση, αναλογική εταιρική σχέση ως προς τις κυρώσεις ή τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο περισσότερο συνεργαστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο θα πριμοδοτηθεί η συνεργασία αυτή και θα ε, διαβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με βάση τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου. Βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι μέλος του κλαμπ. Δεν το επιθυμεί πλέον, το σεβόμαστε ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων δεν θα συμμετέχει στις κοινέ αποφάσεις. Με την εταιρική σχέση όμως αυτή, το Λονδίνο θα είναι ένας από τους δυνατότερους εταίρους μας και θα μας βοηθήσει. Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι στον τρίτο γύρο των πρωτευουσών της Ευρώπης. Κάθε εβδομάδα έρχομαι σε επαφή και με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μακάλιστερ και την Επιτροπή του για την παρακολούθηση του Brexit και τον τρόπο με τον οποίο έχετε συνδράμει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις μελλοντικές μας σχέσεις. Γνωρίζω τις προσδοκίες σας. Εξ αρχής είχα πει ότι δεν διαπραγματευόμαστε θέματα ασφάλειας Θέλουμε να έχουμε μία στεναρή σχέση ως προς την ΚΕΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μία τέτοια όμως εταιρική σχέση χρειάζεται και μία ελάχιστη νομική πλαισίωση και γι' αυτό θέλουμε αυτό το πλαίσιο εξ αρχής, γι' αυτό θα πρέπει να κυρωθεί η συνθήκη αποχώρησης. Διαφορετικά θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες. Δεν επιθυμώ το no deal, την άτακτη αποχώρηση, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει και η άτακτη αποχώρηση στον τομέα της ασφάλειας, δηλαδή μια ρήξη και ε, πλέον μία διαφορετική θεώρηση επί των ζητημάτων ασφαλείας και ανταλλαγής πληροφοριών γιατί οι ανταλλαγές πληροφοριών θα είναι πιο περιορισμένοι. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχει συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις κοινέ επιχειρήσεις, καθώς και ως προς την αμυντική ικανότητα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Η άτακτη αποχώρηση, το no deal, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ενισχυμένη πλαισίωση και κοινή πλαισίωση. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τους στρατηγικούς κινδύνους, όπως είπε και η ύπατη εκπρόσωπος, η Φεντερίκα Μογκερίνη, και θα πρέπει να προωθήσουμε βεβαίως ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, αλλά αυτό θα γίνεται μονομερός και μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Πολύ συχνά είπα ότι λυπάμαι για το Brexit, λυπάμαι για αυτή την έκβαση, ενδεχόμενη έκβαση, αλλά θα ήθελα η αποχώρηση να είναι τακτική είναι μια κατάσταση αμοιβαία απώλειας. Δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία. Είναι μια κατάσταση lose-lose. Όλοι χάνουν. Δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία από το Brexit. Αυτό το καταγράφουμε, λυπούμεθα γι' αυτό και θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα που πρέπει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε γιατί το 52% των Βρετανών αποφάσισε και τάχθηκε κατά της Ευρώπης. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι φόβοι, αυτή η ανασφάλεια και να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες του Brexit και να εισακούμε τους πολίτες. Να υπάρχει μια προστασία, ο Ευρωπαίος πολίτης να νιώθει προστατευμένος. Γι' αυτό θα πρέπει να προτάξουμε μια νέα συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, όποια και να είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν αγαπητέ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Συνάδελφοι, κύριε και κύριοι, έχω έναν πολύ μεγάλο κατάλογο ανθρώπων που θα ήθελα να κάνουν ερωτήσεις. Θα έχω συμφωνήσει με τον κύριο Μπαρινιέ να ακούει τρεις ε, παρεμβάσεις ε, και μετά να απαντά. Τρεις-τρεις λοιπόν θα μιλάνε οι συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω λοιπόν, ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι και ακριβείς για να είμαστε και δίκαιοι και στους άλλους συναδέλφους που περιμένουν να μιλήσουν. Ξεκινάμε με την Βαρόνι Armstrong από το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα σε όλους. Είμαι από την Βουλή των ε, Λόρδων. Αν ε, ήμουν από τη Βουλή των Κοινοτήτων θα είχα άλλες δουλειές. Αλλά Βρίσκομαι εδώ πραγματικά για να συμφωνήσω και με τον κύριο Μπαρνιέλαν και με την έκθεση που βγάλαμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα για τις μελλοντικέ σχέσεις ε, Ηνωμένου Βασιλείου ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέμε πέρα από τον Brexit ε, πώς να κάνετε φίλους και να επηρεάζετε ανθρώπους. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Είναι αρκετά εκτεταμένη η έκθεση και επισημαίνει ότι υπάρχουν τρεις ε, τομείς ε, πέρα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπαρνιέ, κατά μια έννοια, που είναι βασικό στοιχείο των μελλοντικών σχέσεων. Πρώτα απ' όλα, παρά την αβεβαιότητα, για να το πω έτσι, για το τι θα γίνει με την συμφωνία αποχώρησης ότι ο μηχανισμός διακυβέρνησης που περιέχεται στην συμφωνία αυτή μας ε, προσφέρουν μια δομή μελλοντικού διαλόγου που θα παραμείνει και σε οποιαδήποτε συμφωνία καταλήξουμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα πολύ προσεκτικά και με βάση τα όσα είπε ο κύριος Μπαρνιέ αυτό να γίνει κατά τρόπον ώστε θα πηγαίνει πέρα από τις επίσημες δομές για να υπάρχουν επαφές ανθρώπων που ανησυχούν για το μέλλον τους, το οικονομικό τους μέλλον κτλ. για να υπάρχει πραγματικά στήριξη για πραγματική συνεργασία. Δεύτερον, βεβαίως ε, υπάρχουν ε, άλλοι τρόποι, άτυποι αλλά αποτελεσματικοί για την συνεργασία σε τομέα ασφάλειας και για άλλα ζητήματα, ε, καθώς θα είναι μηχανισμοί στους οποίους θα είναι μέλος του ΕΒ και θα πρέπει να έχουμε κάποια σχέση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε και πώς η αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στις ε, Βρυξέλλες ε, θα εργάζεται αποτελεσματικά ακόμα και αν δεν είμαστε μέλος. Ε, αγαπητή Βαρόνη, με συγχωρείτε πρέπει να είμαι αυστηρός με τον χρόνο. Δύο λεπτά, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε. Ε, αυτό το οποίο ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις διεθνώς και έχουμε βρεθεί εδώ λόγω ενός στενού εθνικισμού, πολιτικής ε, ταυτοτήτων και λαϊκισμού. Το δημοψήφισμα έλαβε χώρα κατά διάρκεια της μεταναστευτικής ε, κρίσης ε, και υποφέραμε από αυτό, αλλά το εκμεταλλεύτηκαν και τα άκρα και της δεξιάς και της αριστεράς. Και αυτό το αντιμετωπίζει κάθε χώρα και πρέπει να φροντίσουμε μαζί για να βρούμε τρόπους που θα αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε η δημοκρατία και η συνεργασία να μπορέσουν να ανθίσουν στο μέλλον εντό Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εμεί ήμασταν πολύ φιλικοί με τους Βρετανούς συναδέλφου. Λοιπόν, δύο λεπτά από εδώ και μπρο. Έχουμε λοιπόν πάλι έναν Βρετανό από την Σκωτία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω ξέρετε, οι Σκοτσέζοι είναι λακωνικοί. Λοιπόν, δεν θα βγάλω μεγάλους λόγους. Ε, θα ήθελα και εγώ να σας ε, ευχαριστήσω που διατηρείτε την ε, πειθαρχία. Γενικά είμαι και εγώ λυπημένος για τον Brexit, αλλά βεβαίως νιώθω και αμηχανία για το χάος του Westminster και λυπούμε για το ότι θα υπομένετε αυτούς τους συνομιλητές. Θα τους αντέξετε για λίγο ακόμα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες 24 ώρες η πιθανότερη λύση που προέκυψε είναι η αποχώρηση χωρίς ε, συμφωνία, κάτι το οποίο μας ε, λυπεί. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι είχαμε πει το εάν μπορούμε να δούμε τα δικαιώματα των πολιτών ως μια ξεχωριστή συνθήκη, γιατί πολλοί άνθρωποι βέβαια είναι εχθρικοί σε αυτή τη διαδικασία. Δεν εννοώ την κυρία Μέη, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ε, πραγματικά προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή και θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι ε, να φανούμε πιο μεγαλοψυχοί. Επίσης υπάρχουν οικονομικές πτυχές και άκουσα τις προτάσεις σας για τη δομημένη συνεργασία στην άμυνα, αλλά υπάρχουν και οικονομικές πτυχές για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα μελλοντικά προγράμματα της Ένωσης. Γνωρίζω βέβαια ότι δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα κομισιόν και κράτη-μέλη για τι πτυχέ αυτέ, αλλά μπορείτε ίσω να μα πείτε το τι μπορούμε να περιμένουμε καθώ πηγαίνουμε στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει, ε, εάν φτάσουμε εκεί βεβαίω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρίτος ομιλητής, η κυρία Μπύρο από τη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συνεδρίαση αυτή. Και θα ήθελα βεβαίω ε, να εκφράσω την εκτίμησή μου για την δουλειά που κάνει ο κύριος ε, Μπαρνιέ. Επιτρέψατε μου τώρα να συνεχίσω στην μητρική μου γλώσσα. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι συντεταγμένη και όχι άτακτη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Περιμένουμε συγκεκριμένα μέτρα από το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι είναι και θα είναι σημαντικός μας τέρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει συνεργασία στον τομέα της ΚΕΠΑ, στην άμυνα και ασφάλεια, με βάση τις κοινέ αξίες και προτεραιότητες. Εμείς θα ε, υποστηρίξουμε μία ενισχυμένη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο στα πλαίσια της ΚΕΠ με βάση αυτή την διμερή εταιρική σχέση η οποία θα διαμορφωθεί ανάλογα και με τα επόμενα βήματα του Brexit. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ, για την κυρία Μπυρό πρώτα. Αυτό που λέτε και που εύχεστε για τη χώρα σας, που είναι σε νευραλγική θέση στην ε, περιοχή αυτή της Ευρώπης και που έχει μεγάλη σημασία, δείχνει και τα δεδομένα του προβλήματος, όπως μπορώ να πω και στην ε, Βαρόνι Άμστρομ. Θέλουμε, και αυτό ήταν και το νόημα των λόγων μου έως τώρα, θέλουμε, έχουμε ανάγκη και κοινό συμφέρον να έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε και τα σχετικά συστατικά. Έχουμε το πλαίσιο, χάρη στην πολιτική δήλωση. Άλλωστε αυτό δεν αντιφάσκει με το ότι διμερώς η Ρουμανία, η Γερμανία, η Γαλλία, άλλες χώρες, η Εστονία, η Λιθουανία μπορούν και κάνουν ήδη σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διμερεί συνεργασίε θα συνεχιστούν, είτε επί πολιτικών είτε επί προγραμμάτων. Η συνεργασία εντό του ΝΑΤΟ για τις χώρες εκείνες μέλη της Ένωσης που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, γιατί δεν είναι όλες, θα συνεχιστούν αυτά βεβαίω. Και γι' αυτό και εκφράζουμε ανησυχία για το μέλλον του ΝΑΤΟ. επιθυμεί να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και θα αποχωρήσει. Η παρουσία του ωστόσο, η δυνατότητά του να εκφράζει γνώμη και να συμμετέχει για τις επιχειρήσεις στα προγράμματα και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για την κυρία Άμστρομ, οφείλω να πω την αλήθεια. Δεν είναι το ίδιο με το να είστε μέσα στην Ένωση, εάν είστε έξω. Δεν είναι business as usual, ούτε σε αυτό το τομέα, ούτε και στους υπολείπους. Άρα θα πρέπει να βρεθούν άλλες μορφές και πλαίσια συνεργασίας. Μίλησα ήδη για στρατηγική συνεργασία και μίλησα για τους πέντε μηχανισμούς ε, που επιτρέπουν ε, να συνεχιστεί αυτός ο στρατηγικός και πολιτικός διάλογος. Όμως υπάρχουν, υπάρχουν επιπτώσεις κύριε Άμστρομ. Η χώρα σας αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κοινή αγορά, την Τελωνιακή Ένωση, ως τώρα τουλάχιστον. εγκαταλείπεται με τον τρόπο αυτό. Αποχωρείται και από 750 διεθνείς συμφωνίες. Καλά με ακούσατε. 750 διεθνείς συμφωνίες. Μηχανικά, ε, νομικά. Ε, αποχωρείται από Ευρατόμ, από Ευρωπόλ, από όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Αυτό είναι μια μηχανική, ας πούμε, αυτόματη ε, συνέπεια. Δεν θα επεκταθώ για τα όσα συμβαίνουν το Ηνωμένο Βασίλειο για ένα διέξοδο πολιτικό ή κρίση πολιτική που πάει σε περισσότερο βάθος από το θέμα του Brexit και μόνο. Δεν είναι μονάχα το ζήτημα του Brexit και της συμφωνίας που έχουμε εδώ και του Ιρλανδικού backstop. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος από αυτό. Είναι μια κρίση που μπορεί να υπάρχει και σε άλλες χώρες. Ακούω την κυρία Λιωμαρή ή τον κύριο Μπιζέ και μπορούν να πούν ακούω και για τη χώρα μου, την Γαλλία, σχετικά με το ποια είναι η σχέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο, ποια είναι η θέση μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ποιο ε, πολιτικό μοντέλο θα υιοθετήσουμε. Αυτά όλα θα αναφιούν μέσα από τις συζητήσεις για το Brexit. Εξάλλου, θα συνεχίσω να ε, εκφράζω σεβασμό για τις κοινοβουλευτικέ διαδικασίε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακούω άλλωστε συχνά την κυρία Άμστρομ όταν λαμβάνει το λόγο. Το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ε, συναρπαστική η συζήτηση, αλλά θα συνεχίσω να τηρώ τη δική μου στάση. Εκφράζω τη λύπη μου για το Brexit. Πάντω τη δική μου στάση δεν θα βρείτε ποτέ, ούτε είδατε ποτέ, ούτε θα βρείτε ποτέ οποιαδήποτε διάθεση ταπείνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάντω τώρα έχει έρθει η ώρα να αναλάβετε τι δικέ σα ευθύνε. Και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα αυτό ακριβώ θέλει να πει ανοίγει τον δρόμο ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο για να μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες του. Είτε θα συμφωνήσετε για να μπορέσετε να αποχωρήσετε συντεταγμένα και είναι μόνη δυνατή συμφωνία, διότι την ε, συντάξαμε σε αντικειμενική ε, νομική βάση. Είτε αν δεν θέλετε συμφωνία και αν αποφασίσετε να εξέλθετε χωρίς συμφωνία, αυτό είναι απόφαση δική σας, δική σας ευθύνη, ευθύνη του Ηνωμένου Βασιλείου αν επιθυμεί να αποχωρήσει άνευ συμφωνίας. Ή αλλιώς θα αποφασίσετε να ζητήσετε παράταση. Αλλά θα πρέπει να μας πείτε τότε για ποιο λόγο. Ας πούμε για νέο δημοψήφισμα, για νέες εθνικές εκλογές, για να αναπτυχθεί μια πολιτική διαδικασία διακομματικά. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, εάν τεθεί το θέμα της παρατάσεως, θα, θα ρωτήσουν γιατί. Άλλωστε θα πρέπει να οργανώσετε και ευρωεκλογέ τον Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα αυτό υποχρεωτικό. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω για την ώρα σήμερα. Ε, είπατε και για ε, τις ε, χρηματοδοτικές ρυθμίσεις. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, έτσι δεν είναι. Αν δεν υπάρξει deal. Αυτό δεν εννοείται. Αν υπάρξει συμφωνία, εφαρμόζουμε τις από κοινού υποχρώσεις υποχρεώσει για την προστασία των πολιτών, 4,5 εκατομμύρια πολίτε Και θα υπάρξουν οι ρυθμίσει με τον τρόπο που έχουν προβλεφθεί και θα υπάρξει και μια μετάβαση για μια περίοδο δύο ετών, μέχρι το 2020, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Πρώτα-πρώτα η ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετική, το κλίμα, διότι έλλειψη συμφωνία σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης σημαίνει ε, ρήξη της εμπιστοσύνης. Ενώ εγώ χρειάζομαι, θεωρώ ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη για να χτιστεί ένα κοινό μέλλον. Στην περίπτωση αυτή η χώρα σας θα έχει ανάγκη τις σχέσεις μαζί μας και εμείς μαζί, μαζί τους βέβαια. Δεν θα περάσουν πολλοί μήνες μέχρι ότου το, ευρωπαϊκό, το, το να ζητήσει να ανοίξουν διαπραγματεύσεις για Common Trade Agreement αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στην περίπτωση αυτή τα θέματα του Brexit εξακολουθούν να υπάρχουν. Η Ιρλανδία, οι ε, δημοσιονομικές ρυθμίσεις για την συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα δικαιώματα των πολιτών. Θα ξαναθέσουμε τα θέματα αυτά εάν το Ηνωμένο Βασίλειο επανέλθει να συζητήσει περί εμπορίου, σε περίπτωση no deal δηλαδή, εμπορίου κλπ. Θα τεθούν ξανά τα θέματα αυτά, είναι πραγματικά θέματα. Ε, δικαιώματα των πολιτών, Ιρλανδία, ε, ε, Βρετανική συνεισφορά. Θα ακολουθήσουν τώρα τρεις ευρωβουλευτές, Σαλαφράνκα, Αντζέλ και Φρόιντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΕΛΚ, δηλαδή ότι αναγνωρίζουμε το έργο του βασικού διαπραγματευτή μετά από μεγάλες δυσκολίες και με μεγάλες γεωστρατηγικές απειλές. Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Μπαρνιέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής όχι σε σχέση μόνο με μία ενδεχόμενη συμφωνία, αλλά το εξής. Αυτό που μας απασχολεί είναι τι θα γίνει μέχρι τις 12 Απριλίου. Δηλαδή, αν ε, δεν επιτευχθεί συμφωνία και επέλθει ρήξη, τι θα γίνει με, τα, με το δημοσιονομικό σκέλος αυτής της συμφωνίας ή μη συμφωνίας. Ε, από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να τεθεί επιτάπητος για άλλη μια φορά η συμφωνία. Και εν πάση περιπτώσει όπως έγινε χτες με διαφορά τριών ψήφων, εάν παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Τελωνιακή Ένωση Μισελ, θα πρέπει να γίνει επαναδιαπραγμάτευση ή θα μπορούσαμε να βασιστούμε στην προϋπάρχουσα συμφωνία. Δηλαδή, ο οποιαδήποτε αλλαγή στη συμφωνία σημαίνει επιπρόσθετο χρόνο, τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Ignacio. Σας ευχαριστώ. Ανζέλα, του Λουξεμβούργου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μπαρνιέ, διότι προσέδωσε μεγάλη σημασία στο διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είχε μεταβεί τρεις φορές στο Λουξεμβούργο, γι' αυτό το λόγο και συνομίλησε και με την ε, κοινή γνώμη, με τους πολίτες μας, έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι η Ευρώπη είναι ένα σχέδιο, ένα μεγάλο σχέδιο υπέρ των πολιτών, πέρα από το οικονομικό ή εμπορικό σκέλος και κατανοούν οι πολίτες τι θα χάσουμε αν δεν υπάρχει η Ευρώπη. Βεβαίως, ε, ο τρόπος εργασίας ε, προσέδωσε ενότητα στους 27. Πώς εκτιμάτε τους κινδύνους για το μέλλον όταν θα γίνει η μελλοντική διαπραγμάτευση με το Ηνωμένο Βασίλειο, τι πρέπει να κάνουμε τα προσεχή χρόνια και ως προς τις μελλοντικές μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο έχετε αναγνωρίσει ευαίσθητα στοιχεία που θα μπορούσαν να πλήξουν την ενότητα των 27. Ελπίζω η μέθοδος Μπαρνιέ που είναι η μέθοδος απώλειας, απόλυτης διαφάνειας να αποτελέσει ένα δίδαγμα, μεγάλο δίδαγμα για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Φρόιντ από την Αυστρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω κύριε Μπαρνιέ για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει και όταν ε, ξεκινήσατε φαντάζομαι δεν περιμένατε να είστε εδώ 2 Απριλίου να μας εξηγείτε τι θα είχε συμβεί στις 29 ε, Μαρτίου. Λοιπόν, μετά την δεύτερη ψηφοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο, το είχα πει και το ξαναλέω πριν την πιθανή τέταρτη ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνω πώς ε, είναι απολύτως σαφές και θεμητό να ψηφίζει κανείς τέσσερις φορές για το ίδιο θέμα ε, στο Κοινοβουλίο μέσα σε δύο μήνες, αλλά οι ίδιοι πολιτικοί που φέρνουν τέσσερις φορές το ίδιο νόμο για ψήφισμα αρνούνται να κάνουν ένα δεύτερο δημοψήφισμα τρία χρόνια αργότερα. Ε, ίσως αυτό σχετίζεται με το ότι οι συντηρητικοί φοβούνται πως ε, ε, φοβούνται τι ευρωεκλογέ όπως ο διάολος στον αγιασμό. Γιατί ε, φοβούνται ότι θα επανέλθουν εδώ βουλευτές των εργατικών και θα αυξηθεί έτσι η δύναμη των σοσιαλδημοκρατών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με κάτι τέτοιο ή όχι. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή είναι η τελευταία μου φορά που βρίσκομαι σε συνεδρίαση της Επιτροπής, να σας ευχαριστήσω εσάς, David, για την ε, πολύ καλή και αμερόληπτη δουλειά που έχετε κάνει όσο καιρό είστε πρόεδρος και εύχομαι στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών κάθε επιτυχία και ελπίζω να συνεχίσουν να εργάζονται για μια ισχυρή εξωτερική πολιτική με αυτοπεποίθηση. Σας ευχαριστούμε κύριε Φρόντ. Τελευταία συνεδρίαση πράγματι. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Μίσελ, να ακούσουμε άλλον έναν. Να γίνουν τέσσερις. Να ακούσουμε και μια διαφορετική βρετανική άποψη τώρα. Ο Λόρδος Κίνοκ από τη Βουλή των Λόρδων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κίνολ, με συγχωρείτε. Μου εντύπωση το τι θερμή η υποδοχή είχαμε, γιατί ήμουν επιφυλακτικό ε, κοιτάξτε, είναι πολύ ευαίσθητη η λειτουργία της δημοκρατίας και βλέπουμε το τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μας ε, ε, υπάρχει μία θέση λειτουργία. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να επαναλάβω την άμεση ανάλυση που βλέπετε στο BBC. Μέσω πρόθεσμα, άκουσα προσεκτικά τον κύριο Μπαρνιέ, και σκεφτόμουν η δουλειά απαιτείται μέσω πρόθεσμα για να υπάρξει μια εξέλιξη της ε, σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου όπως την περιέγραψε ο κ. Μπαρνιέ και να εξελιχθεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες ε, που δημιούργησαν αυτό το 52% των ε, Βρετανών που ψήφισαν για να αποχωρήσουμε, γιατί υπάρχουν αυτέ οι ενισχύσεις και σε άλλε χώρε και αν δεν αντιμετωπιστούν θα έχουμε προβλήματα. Θα έχει προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθήσουν και τα εθνικά κοινοβούλια αυτή την εξέλιξη, γιατί βεβαίω οι περισσότερε αποφάσει θα απαιτήσουν ομοφωνία για τι συνθήκε και λέω συνθήκε ε, γιατί θα είναι πολλέ μάλλον από τη, θα προκύψουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν θα είναι θέμα ειδική πλειοψηφία. Μακροπρόθεσμα όμω, ο κοινό στόχο όλων των βουλευτών είναι η ειρήνη και η ευημερία για του εκλογέ του ή στην περίπτωση τη Βουλή των Λονδών για του συμπολίτε μα. Σήμερα χαρήκα που είδα ότι εκπροσωπείται και η Νορβηγία εδώ πέρα Βεβαίω η Νορβηγία δεν είναι κράτο μέλο τη Ένωση και ελπίζω να μας προσκαλείτε και εμά στο μέλλον στι συνεδριάσει αυτέ γιατί εγώ αισθάνομαι πολύ άνετα και πολύ Ευρωπαίος. Ε, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Τσότσιλ ε, συχνά αναφέρεται, αναφέρονται τα λόγια του λάθο, γιατί ε, θεωρούσε ότι βεβαίως το να συνομιλείς είναι ο καλύτερος τρόπος για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Όταν ε, φύγετε, Λόρδε Κίνολ, τη Νορβηγία. Θα ήθελα να πω ότι η Νορβηγία αποφάσισε να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόλο που είχαν τότε γίνει διαπραγματεύσεις προσχώρησης αλλά θεώρησε ότι πρέπει να συμμετάσχει στην ενία αγορά. Και τα πράγματα πάνε πολύ καλά για τη Νορβηγία γιατί η αγορά της δεν είναι εθνική αγορά. Είναι μια αγορά που συνδράμει την Ευρωπαϊκή Ένωση και Τούμπαλιν. Και είχα μία συνάντηση με έναν διπλωμάτη από τη Νορβηγία που είναι κάπου εδώ στην αίθουσα. Τον είχα συναντήσει εδώ και 10 χρόνια και το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα. Λόρδε Κίνολ, Μιλήσατε ε, για τη δυσκολία του όλου διαλόγου με τους Βρετανούς, όπως και ο κύριος Φρόιντ. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτές τις δυσχέρειες. Πολλές φορές οι Βρετανοί μας εκπλήσουν, όπως είπατε κύριε Φρόιντ. Και ίσως να μην έχει λήξει και η όλη διαδικασία έμαθα ότι ίσως γίνει μία άλλη σειρά ενδεικτικών ψηφοφοριών μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Τη στιγμή που υπάρχει μία πιθανότητα μέσα στα πλαίσια του Βρετανικού διαλόγου να αναλάβουν οι Βρετανοί την ευθύνη αυτής της συμφωνίας, τότε θα πρέπει να τους συνδράμουμε. Η κρίση αυτή είναι πολύ σοβαρή, όπως είπα και στην κυρία Armstrong νωρίτερα, και κανείς δεν χαίρεται για την ύπαρξή της. Κανένας δεν χαίρεται για τις εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή. Λόρδε Κίνολ, βεβαίως πρέπει να δείξουμε δυναμισμό αν όλα πάνε καλά θα ανοίξουν νέες διαπραγματεύσεις, ελπίζω το ταχύτερο ε, δυνατόν και είμαστε έτοιμοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις σε όλους τους τομείς που αναγράφονται σε αυτό το ε, κείμενο. Πρόκειται για 12 παράλληλες διαπραγματεύσεις μπορούμε να προτείνουμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την εντολή διαπραγματεύσεων και το ταχύτερο δυνατόν θα ανοίξουμε αυτά τα 12, 10 ή 12 κεφάλαια στο εμπόριο, μεταφορές, συνεργασία αστυνομίας, συνεργασία στο δικαστικό τομέα και ούτω καθεξής. Ε, το διάστημα είναι μικρό, 21 ε, μήνες διαπραγμάτευσης. Μπορεί βέβαια να παραταθεί αυτό το διάστημα, όπως έγινε για την περίπτωση, με την περίπτωση του Καναδά ή της Ιαπωνίας. Και εξάλλου, Λόρδε Κίνολ, και εγώ είπα ε, υπερβαίνοντας κάπως την εντολή του βασικού διαπραγματευτή ότι δεν είναι αργά να αντλήσουμε από τα διδάγματα του Brexit, να ακούσουμε τους πολίτες ε, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία και το θυμό τους. Αυτό είναι ένα θέμα που εντάσσεται, εντάσσεται στις, ε, συζητήσεις που γίνονται ενώπιση των ευρωεκλογών, αλλά και για τα επόμενα ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ανζέλ για την εκτίμησή σας. Ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο. Βεβαίως αυτή η ενότητα δεν ήρθε εξ ουρανού. Διαμορφώθηκε μετά από συμφωνία των αρχηγών κρατών. Είδαμε τι γίνεται με το Brexit Είδαμε ποια είναι η στάση των ΙΠΑ, είδαμε τι συμβαίνει στη Συρία, στη Λιβύη, ποιες είναι και πώς διαμορφώνονται οι επιρροές από την Ρωσία και την Κίνα. Γιατί πέρα από το παρελθόν και πολύ περισσότερο θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί θέλει να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και να μην είναι αλληλέγγυο. Εμείς όμως είμαστε αλληλέγγυοι και θα αλλάξουμε αυτά που πρέπει να αλλάχθουν στην Ευρώπη. Ως προς τη μελλοντική ενότητα, εάν κρατήσουμε αυτή τη μέθοδο που είναι και η κλίδα εμπιστοσύνης, δεν ανησυχώ φυσικά, θα υπάρχουν διχογνωμίες, συζητήσεις, διότι οι 27 χώρες έχουν διαφορετική άποψη. Δεν υπάρχουν τα ίδια οικονομικά ή πολιτισμικά δεδομένα. Άρα, αλλά κύριε Αουζέλ, σημασία έχει η πολιτισμικα δεδομενα αρα αλλα κυριε αγγελ σημασια εχει η ολοκληρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νωρίτερα απάντησα σε έναν δημοσιογράφο από το Sky News μου είπε «Μα δεν είσαστε πολύ αμετάπιστοι, δεν πρέπει να κάνετε και άλλες υποχωρήσεις». Του απάντησα ότι δεν μιλάμε για μια εμπορική συναλλαγή. Δεν μπορούμε να θέσουμε ένα αμφιβόλο την ευρωπαϊκή αγορά και οι Βρετανοί το ξέρουν διότι την συνδημιούργησαν για 44 χρόνια. Γι' αυτό μας τιμούν και μας σέβονται οι πρόεδροι της ε, Κίνας και τον είπα, δεν πρόκειται για μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών. Πρόκειται για ένα σύστημα κοινή ρύθμισης, κανονιστικού πλαισίου και νομικής βάσης. Κοινή νομικής βάσης. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα πόδι μέσα και το άλλο έξω. Αυτό ακριβώς εξηγούσα για δύο χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για ε, τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της Γερμανίας, ε, του Λουξεμβούργου και των άλλων χώρων. Όταν δεν ε, δεχτήκαμε τη συμφωνία Τσέκερς, όπου ελέγχθη ότι ναι, θέλουμε το 25% της αγοράς, δηλαδή τα θετικά, αλλά όχι τα αρνητικά. Δηλαδή θέλουμε ένα 25% της αγοράς και στα υπόλοιπα μπορούμε να αποκλίνουμε. Τους είπαμε όχι, γιατί αυτό δεν ευεργετεί τις επιχειρήσεις μας που τηρούν τους κανόνες. Δεν είναι δογματισμός, είναι μια διαδικασία αποχώρησης. Άρα ε, δεν θα αποδυναμώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή αποχωρούν οι Βρετανοί. Είναι τόσο απλό το ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Σάλα Φράγκα. Απάντησα για τον προϋπολογισμό. Το θέμα αυτό υπάρχει, υφίσταται για οποιασδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τους Βρετανούς, το πρόβλημα παραμένει. Το θέμα της Ιρλανδίας και η δημοσιονομική διευθέτηση. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια νέα βάση εμπιστοσύνης από νομικής πλευράς κάναμε την καλύτερη δυνατή εργασία για αυτή τη συμφωνία, άρα θα τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν θα υπάρχει ε, μίνι συμφωνία. Εάν δεν υπάρχει συνολική συμφωνία, τότε θα υπάρξουν πολλοί κλειδονισμοί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε εμάς, αν και είμαστε έτοιμοι. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε συγκεκριμένα κεφάλαια και ρυθμίσεις. Γι' αυτό δίνω αγώνα μέχρι τέλους. David, ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι η υπομονή των Ευρωπαίων έχει φτάσει στα ωριά της. Εγώ παραμένω ακόμα κάπως υπομονετικός για λίγο, για λίγο καιρό για να δούμε τι θα γίνει. Ίσως αλλάξει η πολιτική δήλωση, ίσως μπορεί να αλλάξει σε λίγες μέρες ή εβδομάδες. Αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη φιλοδοξία γενικότερα. Ελπίζω να μην δυναμητήσουμε την όλη αυτή εργασία μας μέχρι τώρα. Uh, Σε ευχαριστώ, Μισελ. Ενδεικτικές ψηφοφορίες, όπως έλεγε και η αφήσα αυτή η αγγλική του πολέμου. Συνεχίζουμε με ηρεμία. Παρακολουθούμε τις διαδικασίε στην Βουλή των Κοινοτήτων με θαυμασμό. Περνάμε τώρα στου επόμενου τέσσερις ομιλητές. Τέσσερις, εντάξει. Τσάλ Στάνοκ, ο κ. Μπιζέ, ο κ. Νάτ και ο κ. Κόβατς Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μιλώντας εντελώς προσωπικά, γιατί εγώ είμαι μια ε, συντηρητική φιλοευρωπαϊκή μειοψηφία εντός των συντηρητικών για την υπόθεση αυτό. Συμφωνώ μαζί σας ε, κύριε Μισελ. Για μένα το Brexit ήταν μια εγωιστική καταστρεπτική διαδικασία και χωρίς νόημα συμφωνώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει όμως ένα πλεόνασμα ασφαλείας. Είμαστε μέλος του π 5 πυρηνική δύναμη, αποτελεσματικές ενοπλές δυνάμεις, έχουμε ειδική σχέση με τη ΣΥΠΑ, τις σχέσεις με την κοινοπολιτεία, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα της αρχιτεκτονικής αυτής άμυνας και ασφαλείας. Και το να περικοπεί αυτό θα είναι οδυνηρό και πράγματι θα βλάψει και τις δύο πλευρές. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε το κλείσιμο της βάσης ε, για την Αταλάντα στην περιφέρειά μου στο Λονδίνο. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας επιχείρησης υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταπολέμηση της ε, πειρατείας. Τα τελευταία τρία χρόνια λοιπόν λέω πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ στενή συνεργασία ασφαλείας με τους 27 και ε, είπα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καθεστώς ε, παρατηρητού στην Επιτροπή ε, αυτή της ασφάλειας. Καμία από αυτές τις ιδέες δεν πέρασε. Τώρα λοιπόν, μετά τη χθεσινό βραδινή ψηφοφορία, δεν έχουμε καμία ιδέα για το τι θα γίνει με τον Brexit. Ίσως υπάρξει μια νέα ψηφοφορία υπέρ, αλλά δεν ξέρω αν έχει τα κουκιά η κυρία Μέη. Τώρα, κοιτάξτε, Από τις χρησινοβρατινές ψηφοφορίες ε, το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων συγκέντρωσε η εκδοχή του δεύτερου δημοψήφισματος. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τον γκρεμό και στην εξωτερική και στην εσωτερική ασφάλεια. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο απολαμβάνει τα ε, ωφέλη του Eurojust, του χώρου Σέγγεν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Όλα αυτά χάνονται εάν φύγουμε χωρί συμφωνία. Είναι πολύ ευκολότερο να συνεργαστούμε στην ΚΕΠΑ. Τι θα γίνει όμω και με τα θέματα εσωτερική ασφαλείας, Μισελ Μπαρνιέ, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Πώ θα έχουμε πρόσβαση, παραδείγματο χάρη στις βάσεις δεδομένων. Ένα μεγάλο ερώτημα. Σα ευχαριστώ, Τσαλστάνο. Τώρα Ζαμπιζέ από την Γαλλία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα, όπω και πολύ εξημών, να ευχαριστήσω τον Μισελ Μπαρνιέ για την εργασία του και για την ε, στράτευσή του. Και έχω μία ερώτηση σχετικά με μία από τις τελευταίες ενδεικτικές ψηφοφορίες της Βουλής των Κοινοτήτων για την ε, Τελωνιακή Ένωση, η οποία χάθηκε για λίγες ψήφους. Είναι όμως πολύ διαφορετική από τις συμφωνίες της 25ης Νοεμβρίου μεταξύ Τερέζα Μέη και των 27, διότι δεν αναφέρεται στο backstop, δηλαδή στο περίφημο δίχτυ ασφαλείας. Κύριε Μπαργέ, είπατε ότι η ενιαία αγορά που είναι και η πρώτη στον κόσμο είναι κάτι το διαφορετικό γιατί κάνει, ε, έχει συγκεκριμένες αξίες. Εάν θυμηθώ τώρα την 6η Ιουλίου και το σεμινάριο στο Τσέκερς, οι Βρετανοί συναδελφοί μας θεωρούν ότι στη συνέχεια, μετά από την αποχώρησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούν να κάνουν dumping σε διάφορες μορφές και εάν το συνδέσω αυτό με τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικού Εμπορίου κ. Λέσιγκερ που προτείνει στους Βρετανούς εμπορικές σχέσεις 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ε, προϊόντα γεωργικά και διατροφής θα τους αναγκάσει να τροποποιήσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες που τους δεσμεύουν τώρα. Εάν λοιπόν έγινε χθε ψηφοφορία για την Τελωνιακή Ένωση χθε, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 θα δεχόταν ένα θετικό αποτέλεσμα χωρίς ε, το δίκτυο ασφαλείας. Ή θα σήμαινε ότι οι Βρετανοί ε, ε, οδηγούν την Ένωση στο, new, στο no deal που ενδεχομένω θα καταλήξει. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο επόμενος είναι ο Χαβιέρ Νατ. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ. Και εγώ συμμερίζομαι όλες τις ανησυχίες που ακούσαμε από τους προευρωπαϊστές. Αλλά είναι ε, καυκικό το σενάριο σου, ρεαλιστικό. Δηλαδή, πριν πέσει κανείς στο βάραθρο, 12 ημέρες ούτε καν πριν από την έξοδο, επικρατεί το βρετανικό πολιτικό χάος. Μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων, δηλαδή τι γίνεται, είναι σαν ο πνιγμένος να βοηθάει έναν πνιγμένο ένας άλλος κολυμβητής και να τον τραβάει από τα μαλλιά για να τον πνίξει και αυτόν, τον διασώστη δηλαδή. Δεν θα υπάρξει νέα συμφωνία, αλλά θα πρέπει να υπέλθει κάποια συμφωνία πρόκειται για άγνωστους παράγοντες. Αν γίνουν εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποια θα είναι η έκβαση μετά από αυτή τη διετή σύγχυση. Μιλάμε και για ενδεχόμενη παράταση όμως οι Βρετανοί τότε θα πρέπει να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές όπου το 10% των ευρωβουλευτών θα δημιουργήσουν, θα συνδράμουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο έξω. Θα έχουμε Βρετανούς επιτρόπους που επιθυμούν να βρίσκονται εκτός Ένωσης. Είναι ένα οξύμορο, μία αντίφαση και δείχνει ότι αποστέλουμε ένα χαοτικό μήνυμα και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Δηλαδή, για να σώσουμε την τακτική, χάνουμε τη στρατηγική. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Το Brexit θα μπορέσει να συνδράμει και στην κρίση της Σκοτίας και της Ιρλανδίας. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μύρο Κόβατς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Μπαρνί για τη θαυμάσια εργασία που κάνει στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από 50 χρόνια βέβαια, η ηρωνία της ιστορίας είναι αυτή, άλλος Γάλλος, ο στρατηγός Ντεγκόλ, αντιτίθετο στην εισδοχή της Μεγάλης Βρετανίας στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σήμερα έχουμε έναν Γάλλο πάλι ο οποίος διαπραγματεύεται την αποχώρηση της Βρετανίας, στο βάθος όμως της ε, καρδιάς του θα ήθελε η Βρετανία να παραμείνει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή, αυτά τα έχει ιστορία. Θεωρώ αγαπητέ φίλε ότι καλώς κάνετε και τονίζετε το ότι η ιδέα που κρύβεται πίσω από την προσπάθεια αυτή είναι καθαρά να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καταδείξει δηλαδή ότι μπορούν να ζήσουν μια χαρά και χωρί Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξο. Νομίζω ότι, όπως είπε ο Ρωμάνο Πρόντι πριν από λίγε εβδομάδες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και λειτουργεί. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπετε να υπάρχει κίνδυνος ορισμένοι να ακολουθήσουν το μοντέλο του Brexit εάν αποδειχτεί ότι η Μεγάλη Βρετανία μπορεί και λειτουργεί χωρίς την ε, ιδιότητα μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, ε, ευχαριστώ. Μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα γύρο μετά. Ίσως μια-δυο ερωτήσεις, λέει ο κ. Μπανιέ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και ε, ακριβής. Εντυπωσιάστηκα πάντως από τη σύγκριση που άκουσα, διότι όταν έκανα αυτό το νεύμα με τα χέρια μου, ε, χρειάζεται πολύ ταπεινοφροσύνη. Εγώ είμαι ε, βεβαίως στην πολιτική και χάρη στον ε, στρατηγό Ντεγκόλε, αλλά τότε ήμουν 14-15 ετών όταν συνέβησαν τα πράγματα αυτά που λέτε. Άρα ας μην κάνουμε συγκρίσεις που ε, είναι κάπως υπερβολικές, δηλαδή συγκρίνεται το στρατηγό με εμένα. Ε, αν και είμαι μέλος του Γκολικού Κόμματος, λίγα χρόνια μετά την αποχώρηση από την πολιτική του στρατηγού Ντεγκόλε ο ίδιος ο ε, Γάλλος πρόεδρος τότε είχε προτείνει δημοψήφισμα για την ένταξη του ε, Ηνωμένου Βασιλείου και εγώ τότε είχα εκστρατεύσει υπέρ. Δεν θα πω περισσότερα. Πάντως θεωρώ ότι η Ένωση είναι δύναμη. Κύριε Κόβατς, ε, αντικειμενικά θεωρώ ότι ένας αριθμός πολιτικών ηθινόντων σε όλες τις χώρες που ήταν αρχικώς υπέρ τη αποχώρηση της χώρας τους από την ε, Ευρωζώνη, δεν το λένε πλέον αυτό. Αυτό διαπιστώνω. Ωστόσο δεν εξαγάγαμε την διαπραγμάτευση με αυτό το σκοπό. Ε, καμιά διάθεση τιμωρίας ή κακομεταχείρισης των Βρετανών. Όχι, ειλικρινά. Απέφυγα να θέσω οποτεδήποτε ε, κάποιο συναισθηματισμό μέσα στην ε, διαπραγματεύσει αυτή. Κοιτάξαμε μόνο τα νομικά προβλήματα που θέτει το Brexit. Και θα συνεχίσω χωρίς συναισθηματισμούς, χωρίς πάθη. Μιλώ για τα νούμερα και μιλώ για τα αντικειμενικά στοιχεία. Αντικειμενικά όμως, όπως είπε και μέλος της Βουλής των Λόρδων που είναι παρόν εδώ, το γεγονός ότι αποχωρούν από την Τελωνική Ένωση την κοινή αγορά και από 750 διεθνείς συμφωνίες έχει επιπτώσεις. Θα έχει επιπτώσεις. Και ε, τα πράγματα αυτά πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πω επίσης στον Χαβιέρ Νάτ ότι όντω πρέπει να φροντίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπα και πριν. Και είπα μάλιστα κύριε Νάρτ ότι κάθε παράταση, εφόσον ζητηθεί παράταση, θα αναγκάσει το Ηνωμένο Βασίλειο να διεξαγάγει ευρωεκλογέ στην επικράτειά του ε, τον μήνα Μάιο. Και η παράταση θα σημαίνει βέβαια παράταση της αβεβαιότητας. Δηλαδή θα έχει ένα πολιτικό και οικονομικό κόστος. Είναι και ευθύνη μου να του το υπενθυμίσω. Βεβαίω ε, θα είναι υπόθεση και απόφαση των των της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανικής κυβέρνησης. Αν η Βρετανική κυβέρνηση εξηγήσει για ποιο λόγο χρειάζεται την παράταση, και υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι, για παράδειγμα, διεξαγωγή δημοψηφίσματο ή διεξαγωγή νέων εθνικών εκλογών ή ίσω μια νέα πολιτική διαδικασία. Μπορώ να φανταστώ για του λόγου αυτού, ίσω χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Όμω χρόνο που χρειάζονται οι ίδιοι Βρετανοί για να προχωρήσουν την πολιτική του διαδικασία. Πάντω κάθε παράταση έχει ένα κόστο. Πέραν του γεγονότο ότι υπάρχει και αυτό το παράδοξο, δηλαδή όταν κάποιο θέλει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει ταυτόχρονα να είναι και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συνεχίζει να δίνει τη γνώμη του. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το, Ευρωπαϊκό, ε, το, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα παραμένει μέχρι την αποχώρησή του. Ελπίζω και πάλι ότι τις λίγες μέρες που απομένουν θα μπορέσει να βρεθεί ένας δρόμος για να προχωρήσουμε στην έγκριση της ε, συμφωνίας και το άνοιγμα αυτής της πόρτας για να μπορέσουμε να αρχίσουμε το δυνατόν συντομότερο τη νέα διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ και τον Ζαν Μπιζέ μάλλον, για, το, για την κρίση που εξέφρασε. Τώρα, η ψηφοφορία για την Τελωνική Ένωση. Λέω αντικειμενικά ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσει να συμμετέχει στην Τελωνική Ένωση, Τελωνική Ένωση δεν είναι ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Τελωνιακή Ένωση, περνάμε την Τουρκία για παράδειγμα, όπως στην περίπτωση της Τουρκίας θα είναι μια Τουρκία συν, δηλαδή Τουρκία συν αγροτικά προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει μέλος της κοινή μας πολιτικής για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, αλλά δεν θα υπάρχουν πλέον δυνατότητε να διαπραγματεύονται ξεχωριστά με του Αμερικανού παρά μόνο μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και αν δεν υπάρχει η Τελωνιακή Ένωση, ε, αν υπάρχει συμφωνία Free Trade Agreement, ελευθέρων συναλλαγών, θα συζητήσουμε με τους Βρετανούς για ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να αφήσουμε δηλαδή αυτή την ρυθμιστική απόκληση. Κοιτάξτε, ε, κυρίε και κύριοι, συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι κάτι το εξαιρετικό εξαιρετικά νέο. Έχουμε, δεν θα είναι μάλλον, έχουμε τέτοιες συμφωνίες πρόσφατα με τον Καναδά, την Κορέα, την Ιαπωνία. Σε όλες αυτές μιλούμε για ε, ρυθμιστική σύγκληση. Προσεγγίζουμε δηλαδή πρότυπα και προδιαγραφές ώστε να μπορέσουμε να εμπορευτούμε μαζί του καλύτερα. Στην περίπτωση όμω του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι το αντίθετο. Σήμερα είναι απολύτω ενταγμένοι, χάρη στην νέα αγορά, και επιθυμούν να αποκλίνουν. Το ερώτημα είναι αυτή η απόκληση που θα πάει. Θα παραμείνει μέσα σε εύλογα όρια ελεγχόμενη, από ποιον ελεγχόμενη ή θα ανοίξουν οι πόρτες σε μηχανισμούς dumping οικονομικό, ε, κοινωνικό, κατά των καταναλωτών και εναντίον μας βεβαίως. Δεν είμαστε βέβαια και αφελείς. Θα ελέγξουμε την απόκληση αυτή και θα φροντίσουμε να υπάρξει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Για τον ε, φίλο Charles Τάνοκ, τον οποίο γνωρίζω καλά και γνωρίζω τις απόψεις του. Charles, πάλι το μόνο που μπορώ να πω, δυστυχώς δεν είναι business as usual. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες που επιφέρει το Brexit. Για παράδειγμα, να είστε παρατηρητές στην ε, κόψη, στην πίεση δεν θα είναι δυνατόν. Και να μην λησμονήσουμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις σχέσεις μας με άλλες τρίτε χώρε. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Ό,τι δίνουμε δηλαδή σε μία τρίτη χώρα θα πρέπει να μπορέσουμε να το δώσουμε και σε άλλη τρίτη χώρα. Άρα πρέπει να είναι κανείς αρεαλιστή. Βεβαίως και χρειάζεται συμφωνία για να διατηρηθεί μια βάση εμπιστοσύνης αλλά θεωρώ πραγματικά ότι τα όσα έχουμε περιλάβει στην πολιτική δήλωση, οι πέντε μηχανισμοί συνεργασίας, ας μην ψάχνουμε να βρούμε περισσότερα ή ε, να τους αλλάξουμε. Εάν ε, υιοθετήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς σε πνεύμα εμπιστοσύνη και καλή συνεργασία, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Και να διατηρήσουμε και το βρετανικό input, τη βρετανική ε, συνεισφορά στη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής ε, Υπήρου αλλά και στην ακτινοβολία της Ευρωπαϊκής Ένωση προ τα έξω. Είμαι βέβαιο γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχει πάει 11.30 ώρα και ο Επίτροπος Χάν περιμένει ήδη απ' έξω. Ε, λυπούμε, δεν μπορώ να δώσω τον λόγο σε άλλους κατάφερα να καλύψω όλους τους εθνικούς βουλευτές. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Ε, ίσως θα έχετε και άλλη ευκαιρία να μιλήσετε στον Μισελ στην Ολομέλεια στο Στρασβουργό. Τέλος, να πω λίγα λόγια. Μισελ, είναι σημαντικό αυτό για μας. Ότι στο τέλος, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκρίνει τη Συμφωνία Αποχώρησης, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει τον τελικό λόγο θα ψηφίσουμε αν συνενούμε ή όχι και θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή μας επί του θέματος και μετά όταν θα συζητήσουμε τις μελλοντικέ σχέσεις ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο η Επιτροπή μας θα αρχίσει να παίζει τον ρόλο της ως η κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τον καντονισμό. Ε, ούτως ή άλλως είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι. Οπότε σας ευχαριστώ που ήρθατε στη σημερινή συνεδρίαση για την ανταλλαγή αυτή απόψεων και σας ε, ευχαριστώ και σας και την ομάδα σας για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε τα τελευταία χρόνια και υπερασπίζεστε τα συμφέροντά μας. Και αναμένουμε να σας ξαναδούμε. faccio finta di parlare. Order. So, um, may I ask all... Λοιπόν, παρακαλώ τους ε, συναδέλφους που θέλουν να συζητήσουν να να βγουν εκτός της αίθουσας. Κάποιοι εκεί στο βάθος, μπροστά από την εικόνα του κυρίου Ντεγκάσπερη. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο θέμα ορίζω τον κύριο Γιωχάνες Χάν, τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ε, και των διαπραγματεύσεων για την διεύρυνση. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σας καλωσορίζω ιδιαίτερως γιατί πρόκειται για μια επίκαιρη συζήτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα το Κοινοβούλιο ενέκρινε την θέση του για τα μέσα γειτονίας και διεθνούς συνεργασίας και το μέσο πενταξιακής βοήθειας. Στις διαπραγματεύσεις με τα κρατημέλη θα επιμείνουμε στην θέση μας για το ΠΔΠ 2021-2027 ότι θα πρέπει η εξωτερική χρηματοδότηση να χρηματοδοτεί την εξωτερική δράση και να υπάρχει μια πραγματική δημοκρατική αιρεσιμότητα με ρήτρε αναστολής και θα επιμείνουμε στην καταλήμπλοκη του Κοινοβουλίου στην στρατηγική κατεύθυνση των μέσων αυτών. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα για τις συζητήσεις ε, που γίνονται σε σχέση με την πολιτική διεύρυνση. Ε, μας απασχολούν πολύ στην Επιτροπή μας από το 2014 και θα συνεχίσουν βεβαίως να μας απασχολούν, αλλά προτείνω να δώσω λόγο αμέσως στον κύριο Επίτροπο και ελπίζω να έχουμε μετά αρκετό χρόνο για συζήτηση για να καλύψω όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα. Αγαπητέ Ιωάννης, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα μιλήσω γερμανικά. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι και εγώ που έχω την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεύτερον, αντιλαμβάνομαι ότι μόλι τώρα είχατε μία συζήτηση για το Brexit. Δεν ξέρω πόσο έντονη θα είναι και η δική μα συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντική, αλλά βεβαίως όχι τόσο επίγουσα όσο ε, το θέμα της απόφασης ε, στο Westminster. Το χαρτοφυλάκιό μου είναι διπλό, είναι η διεύρυνση και η πολιτική γειτονίας και για τις δύο περιπτώσεις ε, ισχύει το εξή είτε εξάγουμε σταθερότητα είτε εισάγουμε αστάθεια και η αιτιολόγηση βρίσκεται στο ότι και στα Βαλκάνια ή στην γειτονία μας το ε, επίπεδο ζωής είναι σαφώς χαμηλότερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γνωστό παράδειγμα είναι η σχέση μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανία, όπου στην αρχή της δεκαετίας του 1990 το επίπεδο ήταν σχεδόν το ίδιο και σήμερα η Πολωνία είναι με 5 με 6 φορές καλύτερα από την Ουκρανία. Και αυτό είναι το υπόδειγμα το οποίο σε ένα βαθμό έχουμε και στα Βαλκάνια και στη νότια και ανατολική γειτονιά μας. Δηλαδή ο στρατηγικός μας στόχος είναι θα ήθελα να πω ένα όραμα θα έλεγα, να δημιουργήσουμε μια ζώνη ε, ευημερίας ε, έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το χάσμα το οποίο δεν είναι και θετικό, είναι ένα μόνιμο πρόβλημα για εμάς. Ήδη σήμερα στην Ανατολική και Νότια γειτονιά μας ε, έχουμε θα έλεγα γύρω στα 20 εκατομμύρια πρόσφυγες, ε, εσωτερικούς ε, πρόσφυγες που δεν θα παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται και ίσως θα μπορούσαν να πάνε σε άλλες χώρες αν δούμε βέβαια και τις δραματικές εξελίξεις στη Συρία αλλά υπάρχει και η Λιβύη και η Ουκρανία και σε μικρότερο βαθμό Νότιος Κάφκασος όπου ε, ζουν ε, διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι ε, βεβαίως θα ήθελαν να ζουν καλύτερα αλλά βεβαίως κοιτάνε και προς την Ευρώπη αυτήν την ε, ήπια δύναμη όπου το επίπεδο του εισοδήματος, το επίπεδο της ζωής είναι σαφώς ε, καλύτερο και υπάρχουν και όλες αυτές οι ατομικές ελευθερίες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο στρατηγικός μας στόχος είναι να προωθήσουμε αυτές τις οικονομικές εξελίξεις ε, και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η κατάσταση του κράτους δικαίου γιατί ε, η υπόθεση είναι κατ' οποίο βέβαιως ε, επαληθεύεται ότι όσο περισσότερο είμαστε σε θέση να δώσουμε κίνητρα σε διεθνείς επενδυτές να πάνε σε αυτές τις ε, χώρες είτε για να κάνουν εμπόριο είτε ακόμη καλύτερα να ιδρύσουν εκεί πέρα θηγατρικές εταιρείε, τόσο περισσότερο επηρεάζει αυτό την ποιότητα και της δικαιοσύνης γιατί βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διαφανές, επαγγελματικό, το οποίο θα λειτουργεί, ένα σύστημα δικαιοσύνης, ε, το οποίο αποτελεί την βάση για τις διεθνείς επενδυτικές αποφάσεις ε, για να πάνε σε ε, αγορές είτε να εμπορευθούν εκεί πέρα. Αυτές είναι λοιπόν οι βασικές μας αρχές τις οποίες υλοποιούμε με διαφορετική ένταση βεβαίως κάθε φορά μπορούν αυτά να εφαρμοστούν καλύτερα εκεί όπου ο εταίρος είναι ένα δυνητικό μελλοντικό κράτος μέλος γιατί στην διαδικασία αυτή μέχρι να φτάσουμε στις διαπραγματεύσεις και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχουμε την υψηλότερη δυνατότητα άσκησης πίεσης ε, για να διαμορφώσουμε διαδικασίες ε, και να επιφέρουμε μεταρρυθμίσεις. Έχουμε λοιπόν αυτό. Ο δεύτερος μοχλός πίεσης είναι με τις ε, χώρες εκείνες οι οποίες έχουμε μια συμφωνία σύνδεσης ή συμφωνία ελευθέρου εμπορίου όπως η Ουκρανία, Μολαβία, Γεωργία μολδαβια ε, γεωργια συμβαίνει αυτό και μετά σε κάποια διαφορετική μορφή με τους άλλους εταίρους ε, ανάλογα με το είδος ε, της ε, σύμβασης και της συνεργασίας. Συνολικά, για να δω την συνολική εικόνα και θα αναφερθώ τώρα ανά περιοχή, θεωρώ ότι στα Δυτικά Βαλκάνια τα τελευταία χρόνια συνολικά έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Εγώ ζητάω πάντα ένα μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου για να κρίνουμε τα πράγματα γιατί υπάρχουν πάντα και οπισθοχωρήσεις αλλά συνολικά θα έλεγα πως υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την οικονομία, το κράτος δικαίου αλλά βεβαίως και όλα αυτά τα οποία λέμε και θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ως συμφιλίωση. Παράδειγμα Υπάρχει αυτή τη στιγμή βεβαίως μια στασιμότητα στον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνας. Ελπίζω να ξεπεραστεί σύντομα γιατί μια λύση του ζητήματος αυτού και ο στόχος ε, μιας τελικά νομικά δεσμευτικής ε, συμφωνίας ε, μεταξύ των δύο χωρών είναι η βασική προϋπόθεση για την συνολική περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί πολλά περιφερειακά έργα σχετίζονται ε, με την βελτίωση των σχέσεων αλλά όλα αυτά έχει επιτευχθεί ένα επίπεδο που αν προκύψουν κάποια κατά τόπους ε, προβλήματα η φυσική αντίδραση είναι η αρμόδιοι να σηκώσουν το τηλέφωνο να μιλήσουν, ε, να δουν πώς ε, θα καθησυχάσουν ξανά την κατάσταση. Πριν από λίγα χρόνια ίσως κατέληγε σε κάποια βίαιη αντιπαράθεση Οπότε θεωρώ εδώ ότι υπάρχει μια σαφής πρόοδος. Μια άλλη σαφής πρόοδος ε, είναι ε, βασιζόμενη στη στρατηγική μας για τα Δυτικά Βαλκάνια που παρουσιάσαμε πριν από ένα χρόνο ως Κομισιόν και είπαμε ότι θα δεχτούμε ένα νέο κράτος μέλος ε, εάν επιλύσει μια διμερή σύγκρουση ε, και από την εμπειρία των παλαιότερων ε, ε, εντάξεων δεν θέλουμε να εισάγουμε διμερείς συγκρούσεις με ό,τι προβλήματα αυτές έχουν και αυτό οδήγησε τελικά στο ότι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ξομάλλε τη σχέση της με την Βουλγαρία αλλά κυρίως και αυτή την πολυετή μια φορά με την Ελλάδα για το όνομα και τώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς ως ε, Βόρεια Μακεδονία και έτσι ε, είναι πλέον η μόνη χώρα από τις έξι της ε, περιοχής που δεν έχει κάποιο ανοιχτό διμερές θέμα με τους γειτονές της σε αντίθεση με όλες τις άλλες. Αυτό δείχνει λοιπόν την ε, δυναμική που ε, υπάρχει στην διαδικασία αυτή. Επίσης σημαντικό είναι και εδώ πέρα απευθύνομαι κυρίως τους ε, συναδέλφους από τα κράτη-μέλη πρέπει να δούμε τις μακροπρόθεσμες προοπτικές και εμείς ως Κομισιόν τέλος Μαΐου θα υποβάλουμε την ετήσια έκθεση πρόοδου για την κατάσταση της ε, κάθε χώρας στην περιοχή, συν βεβαίως ε, την Τουρκία. Και υποθέτω ότι με βάση τα όσα παρατηρούμε θα κάνουμε μία σύσταση και για την Βορεια και για την Αλβανία να περάσουμε στην ε, προετοιμασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ε, επισήμως. Ιδιαίτερα μετά τις ε, θετικές εξελίξεις στην Βόρειο Μακεδονία μου φαίνεται ότι αυτό είναι λογικό και ήδη πριν από ένα έτος είχαμε μια πάρα πολύ ε, θετική ε, στάση 25-26 κρατών μελών και τώρα έχουμε, ε, έχει επιληθεί και το θέμα αυτό του ονόματος και θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Γιατί θεωρώ ότι είναι γνωστό σε αυτήν την Επιτροπή πως κάθε μέτρο που βασίζεται στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης, αλλά και κάθε βήμα στην ε, διαδικασία της ε, διεύρυνσης ε, χρειάζεται ομοφωνία όλων των κρατών μελών και για κάθε φάση της διαδικασίας ένταξης υπάρχουν κριτήρια υπάρχουν προϋποθέσεις ε, που πρέπει να πληρούν οι εταίροι μας. Και αυτές είναι προϋποθέσεις ε, που κρίνουν ε, ομόφωνα και αποφάσισαν ομόφωνα όλα τα κράτη-μέλη και τελικά τα συμφωνούμε και με τους εταίρους μας. Και είμαι βαθύτατα πεπισμένος πως εάν οι εταίροι μας πληρούν αυτά τα κριτήρια είναι και θέμα μετά δικής μας αξιοπιστίας ε, να ανταποκριθούμε και εμείς. Δηλαδή όταν πληρούν οι εταίροι τα κριτήρια για την έναρξη των συνομιλιών θα πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε θετικά. Αξαρτήτως του ότι σήμερα και εδώ πέρα απευθύνομαι σε κάποιους που ανησυχούν στο ότι μια χύψη χώρα θα μπορούσε να ενταχθεί ε, μεθαύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, με τον τελευταίο κράτος μέλος στην Κροατία διαπραγματευτήκαμε 8 χρόνια και ε, δεν υποθέτω ότι οι διαπραγματεύσεις εντωμεταξύ της λέμε διαδικασίας θα είναι συντομότερες. Το πιθανότερο είναι ότι θα κρατήσουν περισσότερο, αλλά είναι ακριβώς αυτή η χρονική φάση όπου όπως είπα έχουμε την δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση για να αλλάξουμε τα πράγματα. Η εμπειρία από τις προηγούμενες εντάξει ε, μας ε, δείχνει ότι δεν επαρκεί παραδείγματος χάρη πλέον να περνάνε κάποιους νόμους ε, οι εταίροι μας που αποτελούν βεβαίως τη βασική προϋπόθεση αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε και πώς εφαρμόζονται αυτοί σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, όταν υπάρχει παραδείγματος χάρη η καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες αυτές τις χώρες, υπάρχει ένα επαρκές νομικό πλαίσιο. Ε, αλλά το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται αυτό, πόσο αξιόπιστο είναι και πόσο αξιόπιστη είναι και η αλλαγή τη συμπεριφορά ε, του συστήματος τη δικαιοσύνη και τα λοιπά για να υπάρχει έτσι μια εγγύηση στο τέλος της ε, διαδικασίας έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ναι αυτές οι χώρες ε, ανταποκρίνονται στι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Λοιπόν, τα εξηγώ αυτά γιατί μας ασκούν συχνά κριτική ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε το ότι στα Βαλκάνια ε, υπάρχουν άλλες ε, πολιτικές ε, δυνάμεις, δηλαδή η Ρωσία, η Κίνα που δραστηριοποιούνται, αλλά και η Τουρκία, αραβικές χώρες κτλ. Τώρα, λοιπόν, επί της αρχής, στην πολιτική ισχύει πάντα το ότι ο φόβος είναι κακός σύμβουλος, οπότε εγώ θα έλεγα το εξής να δούμε την οικονομική θέση της Ευρώπης ε, στα Βαλκάνια. Ε, είναι αναπόφευκτη η Ευρώπη. 75% του εμπορίου των Βαλκανίων είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 75% των ξένων επενδύσεων είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Παρόλα αυτά, εδώ και εκεί, σε, κάποια, σε κάποιες χώρες, σε κάποια έργα υποδομών, υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν έντονη παρουσία και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορώ. Να, μπορούμε να μιλήσουμε για την χύψη χώρα. Ε, λίγες παρατηρήσεις για την ανατολική γειτονία. Εδώ πέρα σε λίγες εβδομάδες ε, κλείνουμε 10 χρόνια. Έχουμε βρει λοιπόν, θεωρώ, ένα μοντέλο για το πώς ε, θα συμβιβάζουμε τα διαφορετικά συμφέροντα των εταίρων μας και τα δικά μας ε, βεβαίως και αυτό όπως είπα είναι πρώτα απ' όλα τα οικονομικά ζητήματα αλλά και τα θέματα της ε, θεμελίωσης του κράτους δικαίου. Θεωρώ συνολικά λοιπόν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε τώρα αναπτύξει το μοντέλο αυτό των λεγόμενων παραδοτέων, όπου ε, οι χώρες αυτές ε, σταδιακά έρχονται πιο κοντά στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με μια διαδικασία πρόσδεσης. Υπάρχουν, υπάρχει ήδη η πρώτη φάση των παραδοτέων μέχρι το 2020 και κοιτάμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα για την επόμενη δεκαετία και συνολικά Ε, θεωρώ ότι έχουμε μια, πολιτική, μια θετική εξέλιξη. Ε, δυσκολότερη διαφαίνεται η κατάσταση στον ε, Νότο. Ξέρετε, έχουμε διαφορετικά δεδομένα εκεί και με τη συνεργασία με την Τινησία όπου ακριβώς υπάρχει το θέμα της δημοκρατικής διαδικασίας που πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αλλά και να χειριστούμε την κατάσταση έτσι ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες ε, προς ε, την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Ιωάννης, για την εισαγωγή σε θέματα πολιτικής γειτονίας και διεύρυνσης. Έχουμε περίπου 35 λεπτά στη διάθεσή μας για συζήτηση με τον κύριο Επιτροπό. Θα παρακαλέσω και πάλι τους αδέρφους να τοποθετούνται σύντομα, θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όσο δυνατόν περισσότερα πρόσωπα, αρχίζοντας με πόσους θέλετε να ακούσετε κάθε φορά, πόσους αντέχεις Ιωάννης. Θα σημειώνω εγώ, θα σημειώνω. Καλά, αρχίζουμε λοιπόν με την κυρία Ζούιτσα που είναι ε, αναπληρώτης, αντι, μάλλον αντιπρόεδρος μας. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Χαν, όπως ξέρετε παρακολουθώ προσεκτικά τα του χαρτοφυλακίου σας και ιδίω για την Ανατολική γειτονία και ακόμα περισσότερο για θέματα νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα λεγόμενα Δυτικά Βαλκάνια. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την περιοχή αυτή του κόσμου και να μην τους αφήσουμε, να μην αφήσουμε τις χώρες αυτές ε, χωρίς βοήθεια. Υπάρχει πρόοδος, όπως είπατε, ιδιαίτερος ενδιαφέρομαι εγώ για τη Βοσνία ριζεγοβινη όσοι γνωρίζετε προέρχομαι από την Κροατία. Και εκεί έχουμε το μακρότερο χερσαίο σύνορο μεταξύ Κροατίας και Βοσνίας Ερσιγοβίνης και Μαυροβουνίου. Μακρότερο σύνορο και, ανάμεσα, και από αυτό που είναι ανάμεσα Φιλανδία και Ρωσία. Άρα είναι πολύ σημαντικά τα όσα συμβαίνουν εκεί. Μιλήσατε για Ρωσία, Κίνα, Τουρκία και κάποιες άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για το μέρος αυτό του κόσμου και αυτό είναι αλήθεια. Είμαι όμως επίσης βεβαία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο παρούσα εκεί από ποτέ και πρέπει να είμαστε παρόντες. Πρέπει να εμπλεκόμαστε σαφέστατα και σοβαρά με το μέρος αυτού του κόσμου εάν θέλουμε οι χώρες αυτές να είναι μαζί μας. Αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται κάθε φορά προσαρμοσμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια. Έχω μια ερώτηση όμως. Ο, επειδή είμαι υπέρ τη αλλαγή του τρόπου ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. Είπατε ότι θα πρέπει όλα τα benchmark, όλα τα ορόσημα των εισαγωγικών, να έχουν ομόφωνη έγκριση. Αυτό ήταν μάλιστα και στην ημερήσια διάταξή μα σήμερα. Τι θεωρείτε, είναι σωστό ότι ορισμένε χώρε θα μπορούν να προβάλλουν βέτο. Γιατί θα πρέπει να συμβαζόμαστε. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τον τρόπο αλλαγής, μάλλον με την αλλαγή του τρόπου ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Και είναι σωστό να έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες προβάλλουν βέτο και επομένως υπονομεύουν την πρόοδο. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Ευχαριστώ κύριε Ζουίτσα. Από Εθνικό Κοινοβούλιο τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τσίγκλης από την Λιθουανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με απασχολεί περίπου το ίδιο ερώτημα. Δηλαδή του βέτο. Όπως είπατε και στην αρχική σας τοποθέτηση σχετικά με διμερείς συγκρούσεις. Πώς να βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες οι οποίες εμπλέκονται σε διμερείς συγκρούσεις. Κύριε Χάν όμως, η Ουκρανία δεν εμπλέκεται σε διμερή σύγκρουση. Υφίσταται κατοχή τμήματος επικρατείας της από χώρα που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τη Ρωσία. Και η Ουκρανία Μάλλον η σύγκρουση εκεί ξεκίνησε από την ρωσική πλευρά, με την προσάρτηση της Κρυμαίας και τώρα με τις εχθροπραξίες στην Ανατολική Ουκρανία. Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται στην πραγματικότητα για το ποιόν της Ευρωπαϊκής Αλληλικής. Όταν μιλούμε για τον Nord Stream 2 και κάποιες προτεραιότητες σχετικά με τις ε, σχέσεις με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο κλπ. Και από την άλλη μεριά με χώρες όπως η Ουκρανία που μάλιστα προχθές έγιναν και εκλογές εκεί. Μάλιστα ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Και η χώρα αυτή τώρα βήμα προς βήμα προσεγγίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως είναι ασαφές πώς θα συνεχίσουμε αυτή την διεύρυνση προς τα ανατολικά όταν υπάρχει αντίθεση από τη Ρωσία. Στα Βαλκάνια δεν υπάρχει αντίθετη θέση, αλλά η διεύρυνση προς τα ανατολικά πού πηγαίνει. Και τι κάνουμε επομένω. όταν δεν υπάρχει ισορροπία στις σχέσεις μας απέναντι στη Ρωσία, από, που είναι προμηθευτής φυσικού αερίου και έχουμε τον αγωγό Nord Stream 2, ενώ η Ουκρανία συνδέεται με το δικό μας ευρωπαϊκό σύστημα αξιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, ο πρόεδρος. Ε, ως ευρωβουλευτής τώρα ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ κύριε Επίτροπε. Τις μέρες αυτές είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου σας και όσα έχουν συμβεί τα το τελευταίο διάστημα. Η ερώτησή μου έχει ως εξή. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι πολίτες τους δηλαδή, κατεβαίνουν στους δρόμους και διαδηλώνουν κατά των κυβερνήσεων. Ορισμένοι αναλυτές μιλούν μάλιστα για άνοιξη των Βαλκανίων. Από τότε που τελείωσε ο πόλεμος εκεί, οι ε, χώρες αυτές υφίστανται σοβαρές διασπάσεις. Λόγω της έλλειψης προοπτικών, δεκάδες χιλιάδες πολιτών εγκαταλείπουν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, βλέπουμε ταυτόχρονα ε, να γίνεται πιο αργός ο ρυθμός της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, πώς τα εκτιμάτε όλα αυτά. Ποιες είναι οι πιθανότητες για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία να αρχίσουν ενταξιακέ διαπραγματεύσει μετά από το ε, Συμβούλιο του Ιουνίου. Γιατί κάτι τέτοιο θα είναι μια πάρα πολύ καλοδεχούμενη πρόοδο στην περίοδο μετά την Σόφια, όπου πολλοί είχαν σημαντικές προσδοκίες για μια νέα διεύρυνση, προσδοκίες που φαίνεται όμω να έχουν χαθεί, δυστυχώς. Ε, ευχαριστώ κύριε Πίτσουλα και κύριε Μισόφκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με Ρωσία, Τουρκία και Σαουδική Αραβία που έχουν εγκατασταθεί πλέον στη Βοσνία Ζιγοβίνη και με την Κίνα να γίνεται ο μέγας χρηματοδότης εκεί, μπορούν οι Βρυξέλλες να κάνουν κάτι για να επιστρέψουν τον κύριο Ζεμπέτ και για να ρωτήσω ποιε είναι οι απόψει σας για τις τρει κοινότητε που δεν μπορούν να φτιάξουν κυβέρνηση γιατί αυτό είναι ο μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα αυτή και τι γίνεται με την αιρεσιμότητα από την πλευρά ε, των Βοσνίων για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και επίσης με τις ποσοστώσεις για το Υπουργικό Συμβούλιο από τις άλλες εθνότητες εκεί. Πήγα με τους άλλους συναδέλφους μου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βοσνία Ζεγοβίνη μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και διαπίστωσα μεγάλη απογοήτευση από την πλευρά και των τριών κοινοτήτων και των θρησκευτικών ηγετών τους μάλιστα, διότι δεν προχωρούν τα πράγματα. Θα ακολουθήσει ο κ. Τόσκα από την Ελληνική Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2018 ήταν μια πολύ θετική χρονιά για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Ε, όχι μόνο για, την, ε, για τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά έδωσε όθηση η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία δημιούργησε μια νέα ατμόσφαιρα και ένα νέο περιβάλλον. Ε, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για πρώτη φορά μετά από 30 σχεδόν χρόνια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας επισκέπτεται επίσημα ε, τα Σκόπια και εκεί θα συζητηθούν ε, διμερεί θέματα και θα υπογραφούν ε, διμερείς συμφωνίες. Κύριο ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι η δυναμική αυτή να αξιοποιηθεί και να προχωρήσουν τα θέματα της ενταξιακής πορείας ε, των ε, χωρών της ε, περιοχής. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μαύρη τρύπα στην περιοχή. Δεν πρέπει να αφήσουμε την επιρροή τρίτων δυνάμεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, ιδίω εκείνων που αποβλέπουν σε ενίσχυση του Ισλαμικού ριζοσπαστισμού ή που θέλουν να διασπάσουν και να αποδυναμώσουν την Ευρώπη. Αναφέρατε, κύριε Επίτροπε, σωστά ότι πρέπει να προωθηθούν αναπτυξιακά σχέδια στην περιοχή, σχέδια που να έχουν σχέση με την ενέργεια, με τα οικονομικά θέματα, γιατί έτσι θα κρατήσουν τον κόσμο στην περιοχή, θα μειώσουν τη μετανάστευση προς την υπόλοιπη Ευρώπη και θα υπάρξουν καλύτερες συνεργασίες και για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και για το οργανωμένο έγκλημα και για τη ριζοσπαστικοποίηση και για θέματα εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών. Υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχουν και τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν προβλήματα με προσπάθεια των αλβανικών αρχών να κατεδαφίσουν ε, κτίρια, σπίτια των ε, ε, κατοίκων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, κάτι που ευτυχώς ανακλήθηκε. Η Ελλάδα επιθυμεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στο Συμβούλιο του Προσεχούς Ιουνίου, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η Αλβανία θα έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις, ιδίω στα θέματα των μειονοτικών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και των σχέσεων καλής γειτονίας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και στα υπόλοιπα θέματα, όπως είναι οι σχέσεις Βελιγραδίου-Πρίστινας και στα υπόλοιπα θέματα της περιοχής και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις επαφές μας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με άλλες χώρες. Ευχαριστώ προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Thank you, dear colleague. Uh, next is Mr. Kosu. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Οι περισσότεροι μίλησαν για μια στασιμότητα της Ευρωπαϊκής να διευρύνει τα σύνορά της. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέληση σε αυτή την περίοδο κρίσης και λιτότητας να διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί υποψήφοι έχουν κάπως αρνητική στάση πλέον ή στάση παλινοδίας σε σχέση με ενδεχόμενη προσχώρηση. Στην Τουρκία η κατάσταση βρίσκεται σε μια στασιμότητα. Τη στιγμή που η Τουρκία δεν τηρεί τι συμβάσει της Κοπενχάγης δεν μπορούν να ανοιχθούν άλλα κεφάλαια. Η Τουρκία ακολούθησε μια θέση που, ή θέσεις γενικότερα που δεν είναι αποδεκτή σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, ε, Αλβανία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, Σερβία. Υπάρχουν ε, πολλές προκλήσεις το σύστημα δικαιοδοσίας, το δικαστικό σύστημα για να σταματήσει η διαφθορά και υπάρχουν ε, πολλές διενέξεις. στο κοσίφο πεδίο δεν έχει αναγνωριστεί από αρκετές χώρες όπως η Ισπανία και η Σερβία ε, προβάλλει τις αξιώσεις της ε, επί του κοσυφοπεδίου και των μετοχίων και ενισχύει τις σχέσεις ε, με την Ρωσία. Θα αλλάξει κάπως η, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πάταξη της ΝΤΑΕΣ. Ευχαριστούμε η κυρία Μπύρο από την Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ. Στα πλαίσια της ε, Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η ε, Ρουμανία προβάλλει την πολιτική διεύρυνση και θέλουμε να υποστηρίξουμε τις ε, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεών τους. Τα Δυτικά Βαλκάνια κατέχουν στρατηγική, γεωστρατηγική θέση και θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη θέση μας του 2008, δηλαδή η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η ΕΙΕΔ θα πρέπει να προωθήσει τις θέσεις της προς Ανατολάς, γιατί ε, πανηγυρίζουμε τη δέκατη επέτειο από την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις χώρες, με τις ανατολικές χώρες. Αυτό αφορά και την τομεακή συνεργασία με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Μολδαβία, ε, Γεωργία και Ουκρανία έχουμε προωθήσει μια εμπορική σχέση στα πλαίσια της ΕΖΕΣ. Υποστηρίζουμε την ενίσχυση του διεθνούς δικαίου καθώς και την γενικότερη ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σάντρα Κανιέτε είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Χάν για την εξαιρετική συνεργασία σε αυτή μας τη θητεία. Κάθε μήνα είχαμε και από μία συνάντηση και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο για να κατοχυρώσουμε τις πολιτικές μας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία ως προς το εξής. Τη στιγμή που έχει επιληθεί το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, δηλαδή το θέμα της ονομασίας, υπάρχει έλλειψη πολιτικής θέλησης να αρχίσουν πραγματικές διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση. Και θυμάμαι το 2003 όταν στη Θεσσαλονίκη μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή προοπτική στα Δυτικά Βαλκάνια, δεν θα είχε ε, νόημα τώρα να υπαναχωρήσουμε, γιατί τα Δυτικά Βαλκάνια κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες στο μεταξύ, γι' αυτό δεν θα πρέπει να επαναληφθεί το σενάριο του 2003. Η κοινή γνώμη τάσεται κατά της διαπραγμάτευσης από ό,τι φαίνεται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για την τρέχουσα κατάσταση διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας για μια πραγματική ένωση. Υπάρχουν πολιτικές φήμες ότι υπάρχει θέμα εθνικής κυριαρχίας της Λευκορωσίας, ότι απειλείται η εθνική της κυριαρχία. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση της κατάστασης και τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου ως προς τα αποτελέσματα των, στις εκλογές της Ουκρανίας, όχι για τον υποψήφιο που κέρδισε, αλλά επειδή ήταν διαφανείς και δημοκρατικές αυτές οι εκλογές. Αυτό αποτελεί μεγάλο μάθημα για τη Ρωσία και δεν νομίζω ότι ο Πούτιν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Ευχαριστούμε. Σαντρα Κανιέτε. Ε, ε, Γιωχάνες, θέλετε να απαντήσετε. Ο Ζόλτα ναι μετέχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Ντέιβιντ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, κύριε Χάν, γιατί συνοψίζουμε την εργασία των παρελθόντων ετών και την εργασία σας σε αυτό το μίζωνος ε, σημασίας θέμα. Νομίζω ότι Πρέπει να σας συγχαρούμε για την προσωπική σας επιτυχία. Δεύτερον, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δύο πάντα συμμετέχουν για να επιτευχθεί συμφωνία ή συζήτηση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προωθήσει τη διεύρυνση και δεν προωθεί σωστές σχέσεις γειτονίας σε σχέση με τους εταίρους μας. Αυτό είναι και το ερώτημά μου, κύριε Χάν. Πώς βλέπετε, μάλλον πόσο έτοιμη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευρυνθεί. Η βασική μου ανησυχία σχετίζεται με την στάση ορισμένων φιλελευθέρων αριστερών κύκλων. Μιλάνε για μεταρρύθμιση σε πρώτη φάση, να μεταρρυθμίσουμε την Ευρωζώνη και τα πάντα γενικά. Και μετά μπορούμε να λάβουμε υπόψη τη διεύρυνση. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ ανησυχητική και επικίνδυνη προσέγγιση. Είμαι πεπισμένος ότι η διεύρυνση είναι μέρος της μεταρρύθμισης και μέρος της λύσης. Και εάν αναβάλουμε αυτή τη διεύρυνση, όπως, γιατί όπως είπε ο κύριος Γιούγκερ, πέντε χρόνια πριν ότι τα πέντε επόμενα χρόνια δεν θα υπάρξει διεύρυνση, είχε βέβαια δίκιο, αλλά φυσικά αυτό ήταν ένα πολύ αρνητικό μήνυμα. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να προωθήσουμε τις προθέσεις μας προς τις χώρες υποδιεύρυνση ότι τις καλωσορίζουμε, τότε νομίζω ότι θα βρεθούμε σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Και αυτή είναι και η σημαντική μου ερώτηση, κυρία Χάν. Πώς βλέπετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενότητά μας και τη συμφωνία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανταποκριθούμε εμείς στο έργο σας. Ευχαριστούμε η κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, Επίτροπο. Ε, καλώς ήλθατε κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες και το έργο σας ε, στο παρελθόν. Επίσης έχει ένα συμβολισμό που το συζητούμε σήμερα το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων, διότι όπως είπε και άλλος συνάδελφος προηγουμένως, ο Τσίπρας, πρώτος αρχηγός κυβερνήσεως, επισκέπτεται επίσημα τη Βόρεια Μακεδονία από το 1991. Και η, ιστορία πραγματικά γράφεται σήμερα στην περιοχή αυτή του κόσμου. Συγχαίρω λοιπόν και τους δύο πρωθυπουργού των ε, δύο χωρών δηλαδή για την σημερινή τους συνάντηση. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό που λέτε, δηλαδή Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία πρέπει να δουν να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές τους και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Έχω ερώτηση τώρα για το Κόσοβο. Ξέρω ότι κυρίως είναι θέμα εσωτερικών υποθέσεων. παρόλα αυτά είναι και πολιτικό το θέμα και πολιτική απόφαση και μιλώ για, την, για το ανεκπλήρωτο καθήκον των θεσμών μας για την ε, απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων για το Κόσοβο. Ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις το Κόσοβο. Η Κομισιόν το είπε πέρσι, το Κοινοβούλιο το δέχτηκε, αλλά η υπόθεση είναι στα χέρια των κυβερνήσεων τώρα. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση των Κοσοβάρων. Δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε ακόμα την ελευθερία θεωρήσεων. Μπορείτε να μας πείτε αν το θέμα αυτό πρόκειται να συζητηθεί και αν θα προσπαθήσετε να επιτύχετε να μπει στην ημερήσια διάταξη της ε, διάσκεψης κορυφής. Και τέλος, η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει χαρτοφυλάκιο διεύρυνσης. Ο κύριος Πέτερλε, Σλοβενία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι σήμερα είναι μια ε, εξαιρετική ημέρα Μιλήσαμε ταυτόχρονα για το Brexit, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, και για τη διεύρυνση. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που είναι κοντά μας σήμερα συνάδελφοι από τις Εθνικές Βουλές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Χάν για την εργασία του και ιδίω για τη συμμετοχή του στην προσπάθεια επίλυσης των πιο σοβαρών και δύσκολων προβλημάτων. Σήμερα η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού γίνεται στην Βόρεια Μακεδονία. Καλό σημάδι αυτό. Και είμαι επίση πολύ ικανοποιημένο για τι καθαρέ θέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ε, διαπραγματεύσει για ένταξη. Για διεύρυνση δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλο χρόνο για να χαθεί. Τώρα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν τα εργαστήρια, τα workshop. Αυτό είναι σημαντικό για όλη αυτή την περιοχή. Και επίση θα συμβάλλει στην σταθερότητα και ειρήνη στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαπραγματεύσει είναι ο καλύτερο δρόμο για να υπάρξει μεταρρύθμιση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Βρετανική αποχώρηση, εδώ συμφωνούμε όλοι. Ελπίζω το ίδιο σύμφωνοι και ενωμένοι να είμαστε και όταν θα επιτεθεί θέμα διεύρυνση με τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πέτερλε. Κόβατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χάν για την ε, πολύ σημαντική τοποθέτησή σας και την έκθεσή σας. Μία σύντομη διευκρίνηση. Η Κροατία διαπραγματεύτηκε μόλις πέντε χρόνια και εννέα μήνες. Χρειάστηκε όμως να περάσει κάποιο διάστημα μετά για την κύρωση. Πέντε χρόνια και εννέα μήνες, ξαναλέω. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν διμερείς διαφορίες, διαφορές ή συγκρούσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο για το Κόσοβο. Και γι' αυτό πολύ σύντομα. Ερώτηση. Ποια είναι η προσωπική σας γνώμη σχετικά με τη δυνατότητα μια ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου. Θεωρείται ότι είναι ρεαλιστική μια τέτοια προοπτική. Και σύντομο σχόλιο. Ανταλλαγή εδαφών υπήρξε μεταξύ, μεταξύ Ανατολικής τότε Γερμανίας και Δυτικού Βερολίνου το 1988. Ε, τι σκέπτεστε λοιπόν σχετικά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορεί να επιτρέψει έτσι την λύση τη ε, διαφορά αυτή και να οδηγήσει σε αμοιβαία αναγνώριση. Ευχαριστώ αγαπητέ Χαν. Έχουμε τώρα, ε, βέβαια το ζήτημα είναι πόσο ακόμα θα έχουμε στη διάθεσή μας τους διερμηνείς, 12.30 λίγη το ωράριο. Έχω ακόμα έξι που θέλουν να λάβουν το λόγο και βέβαια πρέπει να απαντήσει και ο Επίτροπος. Νομίζω εδώ να κάνουμε μια τομή, ας πούμε, να, βάλουμε ε, μια γραμμή για να μπορέσει να μιλήσει ο Επίτροπος. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Έχω πει πάντοτε ότι στην εξωτερική πολιτική θα πρέπει να καταλήγουμε τουλάχιστον σε ενισχυμένες πλειοψηφίες. Κατά βάση, διότι εάν χρειάζεται κάθε φορά η ομοφωνία των 27, 28 και 29, δεν ξέρω τι, τότε είναι σαφές θα είμαστε πάντοτε, ε, θα έχουμε πάντοτε την ικανότητα όχι να δρούμε, αυτό βέβαια να αντιδρούμε σε ό,τι συμβαίνει. Μέχρι την ένταξη χρειαζόμαστε περίπου 300 αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι όλες λιμένες ομόφωνα. Από αυτές τις 300 αποφάσεις, εμένα μου φαίνεται ότι 298 δεν χρειάζεται να ληφθούν ομόφωνα. Είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι η τελική απόφαση για το αν μια χώρα θα πρέπει να γίνει μέλο θα πρέπει να βασίζεται σε μια ομόφωνη απόφαση όλων των χωρών μελών που θα είναι παρούσε σε εκείνη τη στιγμή, που θα είναι δηλαδή μέλη τη Ένωση εκείνη τη στιγμή. Διότι πρόκειται για σοβαρό θέμα αν θα μεγαλώσει η ευρωπαϊκή οικογένεια ή όχι αλλά για την υπόλοιπη ε, διαδικασία ανάμεσα στην αρχή των διαπραγματεύσεων που πρέπει επίσης να είναι ομόφωνη μέχρι το τέλος, δεν χρειάζεται να ισχύει η ομοφωνία. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο και δυνατόν να ισχύσει τουλάχιστον μια ειδική πλειοψηφία. Η ομάδα μου και εγώ περνούμε το 25 μέχρι 30% της, ε, του χρόνου μας και των προσπαθειών μας για να πείσουμε κάποια χώρα μέλος για να στηρίξει μια απόφαση που όλες οι άλλες τη στηρίζουν ούτως ή άλλως από την αρχή. Αυτό είναι βέβαια σε βάρος της αποτελεσματικότητας. Σε ό,τι αφορά τώρα διμερείς συγκρούσεις, μιλήσατε για την Ουκρανία. Εμείς μιλούμε όμως τώρα για, τα Δυτικά Βαλκάνια, δεν μιλούμε για άλλες χώρες. Ε, αυτές οι άλλες χώρες δεν είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Τώρα για το Nord Stream υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ότι δηλαδή για στρατηγικούς λόγους δεν μας ικανοποιεί. Αλλά εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες του κράτους δικαίου. Εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες, τότε είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχθούμε το έργο αυτό υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρούνται, όπως είπα, όλες οι σχετικές διατάξεις. Για τον κύριο Πίτσουλα θα ήμουν προσεκτικός με την χρήση του όρου άνοιξη των Βαλκανίων, διότι οι διαδηλώσεις σε Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία όλες ξεκινούν από διαφορετικές αιτίες και έχουν έντονο εσωτερικό πολιτικό χαρακτήρα και προέρχονται από δυσαρέσκεια απέναντι ε, στα πρόσωπα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Και είναι ε, ειδικό ο χαρακτήρα των ε, εκδηλώσεων αυτών σε κάθε μια από αυτέ τι χώρε. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει κάποιο κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των κινητοποιήσεων. Τώρα, τονίζω και πάλι, όπω είπατε και ορισμένοι εξημών, ότι είμαι πολύ υπέρ και για τη Βόρεια Μακεδονία και για την Αλβανία μετά να αρχίσουμε τις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις. Και για όλους εκείνους που ανησυχούν από την σκέψη αυτή, ξαναλέω ότι η τελική απόφαση, η απόφαση αυτή μάλλον θα σημάνει ότι αρχίζουμε την διαπραγμάτευση Κάνουμε δηλαδή την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πρώτο κεφάλαιο. Και θα ακολουθήσουν αποφάσεις από όλες τις χώρε μέλη. Σχετικά δηλαδή με το ποιο είναι, ποια είναι τα κριτήρια έναρξης των διαπραγματεύσεων για το πρώτο κεφάλαιο. Αλλά πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αν δηλαδή υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους οι χώρες αυτές, τότε είναι ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας και εν τέλει και το να διατηρήσουμε την πολιτική μας μόχλευση στην περιοχή αυτή. Είμαστε οι μόνοι στην περιοχή αυτή που ζητούμε κάτι από τους εταίρους μας. Μόνο εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούμε να κάνουν κάτι. Όλοι οι άλλοι πάνε και τους χαρίζουν εντό εισαγωγικών. Να μην έχουν την εντύπωση όμω, ωστόσο, ότι όλε οι προσπάθειέ του είναι εισμάτιν, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μα δίνει, λένε τώρα, την ελευθερία των προξενικών θεωρήσεων κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν, με την έννοια αυτή, να ανοίξουμε τι διαδικασίε. Γιατί η Βοσνία Ζεγοβίνη, επί του παρόντο δεν εντάσσεται στη διαδικασία αυτή μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εκεί. Ελπίζω τώρα ότι θα μπορέσει να κλείσει η πρώτη φάση με την γνωμοδότηση opinion της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποβληθεί στις χώρες μέλη και ότι μετά θα τη χορηγηθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας που θα ήταν το επόμενο βήμα. Αυτό σημαίνει όμως ότι και οι ηθήνοντες της χώρας αυτής θα καταφέρουν να φτιάξουν κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε, πώς να πω, οι νοσηλευτέ οι οποίοι θα κρατάμε το χεράκι της σα κυβέρνηση. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Έχουν παγώσει για την ώρα οι ενταξιακές βοήθειες. Μάλλον έχουν προσαρμοστεί στην κατάσταση. Και αναμένουμε από την Τουρκία να ενισχύσει την, τις, τους δημοκρατικούς θεσμούς. Τώρα, για τη Ρωσία. Ένα από τα θέματα τώρα λέμε ότι κάθε μια από τις χώρες οι οποίες επιθυμούν να εισέλθουν θα πρέπει να πληρεί απολύτως τα αυτά που αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Συρία. Εμείς τονίσαμε πάντοτε και πρόσφατα σε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Είπαμε ότι επιδιώκουμε πολιτική λύση. Χωρίς πολιτική λύση δεν μπορεί να υπάρξει από μέρους μας υποστήριξη για την ανοικοδόμηση. Και η πολιτική λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει και λύση για την προσωπική ασφάλεια και την ασφάλεια της ιδιοκτησίας και όσων σύρων βρίσκονται ως πρόσφυγες τώρα στην Αλοδαπή. Διότι υπάρχει η ανησυχία ότι πολλοί από τους πρόσφυγες αυτούς, εφόσον επιστρέψουν στην Συρία, θα συλληφθούν από το καθεστώς Άσαντ. Και εν τω μεταξύ έχουν υπάρξει και de facto απαλωτριώσεις ή δημεύσεις των περιουσιών τους. Γι' αυτό πρέπει να λυθούν πρώτα όλα αυτά πριν δώσουμε οποιαδήποτε υποστήριξη. Πάντως μόλις έληξε επιτυχώς η διάσκεψη για τη Συρία που προβλέπει ενίσχυση και για τις πληττόμενε γειτονικέ χώρες της Συρίας, ιδίω η Ορδανία, Λίβανο, αλλά, αλλά εν μέρη και η Τουρκία. Για την κυρία Καρνιέτε. Αυτά που θα κρυθούν να αποφασίσουν οι χώρες μας το καλοκαίρι θα είναι και το απόλυτο τεστ για την ίδια τη δική μας την αξιοπιστία. Αυτό το έχω τονίσει και προηγουμένως. Λευκορωσία. Είναι ένα από τα παραδείγματα εκείνα όπου εδώ και μήνες κολλάει το θέμα σε μια από τις χώρες μέλους για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση των σχέσεων. Δηλαδή προτεραιότητες συνεργασίας με την Λευκορωσία, κάτι που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε πιο εντατικέ σχέσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα η Λευκορωσία να τοποθετηθεί πιο ουδέτερα και να είναι λιγότερο εξαρτημένη. Δεν μιλούμε για να γίνει μέλος της Ένωσης, έχει όμως θεμητό συμφέρον να μπορεί να εμφανιστεί ως ανεξάρτητη χώρα. Και με την έννοια αυτή πρέπει και εμείς να τα αποκριθούμε. Αυτό θα αποτελέσει και προϋπόθεση για περαιτέρω εντατικότερη συνεργασία. Για τον κύριο Νέμετ, αν είμαστε έτοιμοι για διεύρυνση. Νομίζω σε όλες τις χώρες μέλη, αλλά με διαφορετικό βαθμό, θα πρέπει να κάνουμε σχετική προσπάθεια διαφώτισης και ενημέρωση των πολιτών για να κατανοήσουν οι πολίτες για ποιο λόγο το κάνουμε. Επί του παρόντος, πολλοί ηθήνοντες το αντιλαμβάνονται. Όμω ίσω δεν το αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία των πολιτών. Και αυτό είναι επίση σημαντικό να το αντιληφθούν και αυτοί δηλαδή. Κατανοώ την κριτική που ασκούν ορισμένοι, όπω για παράδειγμα ο πρόεδρο Μακρόν, ότι δηλαδή πρώτα πρέπει να εμβαθύνουμε θεσμικά, για παράδειγμα και με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Εγώ νομίζω ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να συμβαδίζουν εκ παραλίλου, διότι και η θεσμική εξέλιξη θα χρειαστεί κάποια χρόνια, αλλά και οι επόμενε διευρύνσει θα χρειαστούν κάποια χρόνια. Αν πω τώρα, πρώτα θα ολοκληρώσω το θεσμικό οικοδόμημα και μετά θα αρχίσω να ασχολούμαι με τη διεύρυνση, τότε χάνουμε όλη αυτή την φόρα που έχουμε πάρει και όλη, όλη το σχεδιασμό και μην λησμονούμε ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που δεν είναι ήδη μέλη μας, συνορεύουν με χώρες που είναι ήδη μέλη της Ένωσης. Στην ουσία πρόκειται για μια συμπλήρωση και όχι διεύρυνση. Για το Κόσοβο τώρα, κυρία Φαγιόν, εκφράζω την ελπίδα ότι οι χώρες μέλη μας, όπως έχω ξαναπεί άλλωστε, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι Κωσοβάροι είχαν να αντιμετωπίσουν 94 κριτήρια και τελικώς τα εκπλήρωσαν όλα. Είναι μια πραγματική σημαντική προσπάθεια. Μεταξύ αυτών ήταν και η λύση διμερών διαφορών. Και εκεί λοιπόν έκαναν σημαντική προσπάθεια. Και μπορώ να πω ότι οι Κωσοβάροι και οι πολιτικοί τους ηθήνοντες και διακομματικά μάλιστα κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι Κωσοβάροι δεν υποβάλλουν αδικαιολόγητες αιτήσει ασύλου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι από τους πιο επιτυχημένους. Έπεισαν δηλαδή τους πολίτες τους ότι κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα. Και αυτό οφείλει να το αναγνωρίσει Και τέλος, land swap, ανταλλαγή εδαφών, δια, διαπραγματεύσει μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Νομίζω ότι θα πρέπει κανεί να τους αφήσει πρώτα-πρώτα στην ησυχία τους να διαπραγματευτούν. Η η συμφωνία μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Αθηνών χρειάστηκε διάστημα και χρειάζεται και 35 σελίδες συμφωνία υποθέτω ότι και μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου θα χρειαστεί παρόμοια προσπάθεια. Αλλά όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το έχω ξαναπεί αυτό, θα πρέπει να οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνευση σε ολόκληρη την περιοχή. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει λύση που να γίνει δεχτή από την ευρωπαϊκή και από τη διεθνή κοινότητα, που ωστόσο να οδηγεί σε ζημία τρίτων. Πρέπει λοιπόν μέσα σε αυτέ τι παραμέτρους να διεξαρθούν οι διαπραγματεύσεις και να ζητηθούν οι λύσει. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, Ιωάννη. Συνάδελφοι, 12 και 35 και ε, η διερμηνία θα τελειώσει σε λίγα λεπτά. σα ευχαριστώ λοιπόν κύριε Επίτροπε για το ότι έχετε κάνει επιτυχημένη υπόθεση την διεύνηση, προωθείτε την δημοκρατία. Λοιπόν, συνάδελφοι, ολοκληρώνεται έτσι η συνεδρίασή μας. Ε, ακολουθεί επίσημο γεύμα για τους Προέδρους Επιτροπών και Επικεφαλής Αντιπροσωπιών στην τραπεζαρία του Προέδρου. Θα σας πούν που είναι οι κλητήρες πριν τελειώσει η συνεδρίασή μας που είναι τελευταία πριν τις ευρωεκλογέ, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που ήρθαν σήμερα συνεδρες, στην συνεδρίασή μας και για τη συνεργασία που είχαμε και αναμένω να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Αλλά για τη συνεδρίαση ευχαριστώ.